Good afternoon, colleagues. Um, we will begin this morning's proceedings with the adoption of the agenda. If there are no objections to the agenda. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με την μερίσια διάταξη. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, εγκρίνετε. Με Κάποιες γρήγορες ανακοινώσεις, πρώτα απ' όλα για τα γλωσσικά. Δεν υπάρχουν κροατικά και γαλλικά σήμερα. Επίσης, η Ανιμπάν, μέλος αυτής της Επιτροπής, ε, είναι σήμερα για τελευταία φορά σε αυτήν την ε, Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να την ευχαριστήσω δημοσίως ε, για τη δουλειά που έχει κάνει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Και να σας πω κάτι άλλο. Για τα νούμερα, ξέρω πως ήσασταν παρόντες στο Στρασβούργο και σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας σήμερα, αλλά καλό ήταν το ότι ήρθατε για να ακούσουμε την Προεδρία. Να πω πως ε, την προηγούμενη φορά είπα πως είχαμε μεγάλο αριθμό τριμερών διαλόγων που ολοκληρώθηκαν ή ε, είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Αυτό πράγματι ισχύει, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής ε, παρέστησαν σε, στο ισοδύναμο 40 συνεδριάσεων. Κάναμε περισσότερη δουλειά από οποιαδήποτε άλλη επιτροπή με ψηλότερη προσέλευση από οποιαδήποτε άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους γιατί κάνετε πολύ καλή δουλειά. Ε, δεν είναι θέμα τώρα του ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά είμαστε οι καλύτεροι. Αλλά το θέμα είναι ότι είδαμε πολλούς ε, παλιούς φίλους ενώ δηλαδή νομοθετήματα τα οποία δεν είχαν προχωρήσει και τα προχωράμε τώρα με τη βοήθεια της γραμματείας την οποία οφείλω να βοηθήσω αλλά και με την βοήθεια των σκιωδών συγητών, των βουλευτών και των βουλευτών βεβαίως που εργάζονται πολύ ενεργά και όλα αυτά βεβαίω υπό την πίεση των εξωτερικών γεγονότων, του προσφυγικού και των άλλων προβλημάτων ασφαλείας που έχουμε και στα οποία έπρεπε να αντιδράσουμε. Οπότε είναι ένα τεράστιο επίτευγμα αυτό το οποίο κάναμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επιπλέον όπως είπα η δουλειά μας ε, συνεχίστηκε εντατικά και σας ευχαριστώ και το λέω γιατί ε, να το πω τώρα γιατί στο τέλος συνεδρίασης θα έχετε φύγει όλοι οπότε περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα τα συμπεράσματα της ε, Λουξεμβουργιανής Προεδρίας δεν θα ξεκινήσω πάλι με τα τυπικά. Όσοι εμπλέκονται σε διαλόγους ε, με την Προεδρία, το ξέρουν. Κάποιος μου εξήγησε ότι εσείς μου το είπατε Ετιέν, ότι η Προεδρία σας είναι ένα συνεχές ε, συμβόλαιο δικαιοσύνης ε, και εσωτερικών. Σιγά σιγά λοιπόν νομίζω και με πολύ σκληρή δουλειά σας από μια μικρή χώρα βέβαια εργαστήκατε πάρα πολύ σκληρά στο νομοθετικό πρόγραμμα αλλά αντιδράσατε και σε κάποια από τα δυσκολότερα ζητήματα που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας τα πείτε λοιπόν και θα τα συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Έτχεν Σνάιντερ, αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας και τον κύριο Ζαν Άσελμπορν, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και βέβαια τον κύριο Φελίξ Μπράζ, Υπουργό Δικαιοσύνης. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά, Ζαν, εσείς θα φύγετε πρώτος, οπότε θα ακούσουμε πρώτον εσάς θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις στα ζητήματα αυτά και μετά θα ακούσουμε τους δύο άλλους υπουργούς. Ξέρω πως έχετε ε, σημαντικά συμβούλια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο κύριος Σουζάν Άσελμπορν, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ από την αρχή της Προεδρίας μας το γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική κρίση. Δράμα, τα συνέχιση των μεταναστευτικών ρευμάτων χωρίς προηγούμενο. Αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, έπρεπε να δράσουμε άμεσα Πραγματικά δημιουργήσαμε, βάλαμε τα θεμέλια θα έλεγα μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, υποδοχή εγκατάσταση, επιλογής και επαναπροώθηση, αν αυτό είναι απαραίτητο. Έλεγχος λοιπόν στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της Ένωσης δείχνει νομίζω ότι η απάντησή μας στην περιπλοκότητα της κατάστασης πάντα σεβόμεθα τις βασικές αρχές της Ένωσης, την αλληλεγγύη, τη φιλοξενία και χρειάστηκε τις αξίες αυτές να τις μεταφράσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Στον τομέα της αλληλεγγύης νομίζω ότι στα πλαίσια της διεθνούς προστασίας προσπαθήσαμε να βρούμε μια συμφωνία για το θέμα της ε, επαναγκατάστασης των ανθρώπων αυτών ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης, αλλά χάρη στη στενή συνεργασία και μαζί σας, και θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, καταφέραμε να ε, επανεγκαταστήσουμε 165.000 και άλλες 20.000 ε, έχουμε βέβαια τώρα μπροστά μας ε, το πρόβλημα της εφαρμογής. Γνωρίζουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι ανεπαρκή και χρειάζεται μεγαλύτερη επιμονή και υπομονή. Για τα hot spots, τα κέντρα επιλογής. Στην αρχή ήταν λίγο αφηρημένη η έννοια αυτή και εδώ και έξι μήνες όταν ξεκινήσαμε, σήμερα όμως είναι πολύ λειτουργικά και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν στον τομέα των hot spots, αλλά έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος. Διαπίστωσα μόνος μου επιτόπου αυτό το οποίο γίνεται. Ε, αυτό που είναι απαράδεκτο είναι ότι κάποιοι δεν θέλουν να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και αυτό θα αμφισβητήσει τις ιδέες που έχουμε συμφωνήσει. Για την επανεγκατάσταση είναι κάτι το οποίο είχαν εξερευνήσει σε εθνικό επίπεδο διάφορες χώρες, τώρα όμως 28 χώρες και συνδεόμενες χώρες όπως η Ελβετία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν αναζητούν να συνεργαστούν μαζί μας. Τα προγράμματα αυτά όπως της επανεγκατάστασης θα πρέπει στο μέλλον να, να αντιπροσωπεύουν θα έλεγα τον κανονικό τρόπο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για τους ανθρώπους αυτούς ε, και ιδιαίτερα για να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας σαν χώρες που υποδεχόμαστε τους περισσότερους πρόσφυγες στον κόσμο. Έχει ξεκινήσει και ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα για την Τουρκία. Δεν θα πρέπει εδώ να δημιουργηθούν προσδοκίες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Νομίζω όμως ότι οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί ε, θα είναι ανταλλάξιμες θα υπάρξει περαιτέρω αλληλεγγύη με τις τρίτες χώρες, μιλάμε για παγκόσμια σφαιρική κρίση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις αιτίες της. Ε, κάποιες χώρες ε, υφίστανται πολύ σκληρές ε, θα έλεγα επιβαρύνσεις και απαιτούν να υπάρξουν λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε και την οικονομική, υλική και λειτουργική συνεργασία της με τρίτες χώρες, παράλληλα με την προσπάθεια η οποία έχει γίνει στα πλαίσια των υπαρχουσών μορφών συνεργασίας τους τελευταίους έξι μήνες συνεργαστήκαμε και με χώρες ε, της Αφρικής, ε, συνάντηση κορυφής ε, της Βαλέτα και επίσης υπογράψαμε και τη συμφωνία για την κινητικότητα με την Αιθιοπία, με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με την Τουρκία. Θυμίζω τη συνάντηση που έγινε για τη μεταναστευτική ροή στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η συνεργασία όμως θα πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι τα προγράμματα δράσης που συμφωνήθηκαν δεν θα πρέπει να παραμείνουν γράμμα νεκρό. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν με συγκεκριμένο τρόπο και να υπάρξει σωστή εποπτεία τους έτσι ώστε να καλύψουμε τις τοπικές επιπτώσεις. Σε επίπεδο ευθυνών εμείς πρέπει να υποδεχθούμε αυτούς που έχουν ανάγκη προστασίας, θα πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και δυστυχώς θα πρέπει να επαναπροωθήσουμε αυτούς που δεν θα πρέπει να τύχουν διεθνούς προστασίας. Για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό της άτακτης αν θέλετε μετανάστευσης πρέπει να ενθαρρυνθεί η νόμιμη μετανάστευση. Οι πολιτικές μας θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και θα πρέπει να συνοδεύονται και από αποτελεσματικές πολιτικές επαναπροώθησης, ιδιαίτερα κάτω από την πίεση την οποία εφιστάμεθα σήμερα. Γι' αυτό η Προεδρία του Λουξεμβούργου έχει υιοθετήσει λειτουργικά στοχευμένες δράσεις για μια τέτοια πολιτική. Θα πρέπει να αποφύγουμε μέσω των hot spot στην Ιταλία και στην Ελλάδα να δημιουργηθεί μια, ένα συνοστισμός αν θέλετε των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν μπορεί να αποχωρήσουν άμεσα. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε μέσω των πολιτικών μας να βρεθούν λύσεις. Ε, στο πλαίσιο αυτό και η αναθεώρηση της ενταλής του Frontex θα παίξει ε, καθοριστικό ρόλο και χαιρετώ εδώ την προ... χαιρετίζω συγγνώμη, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της προηγούμενης εβδομάδας. Βραχυπρόθεσμα εμείς ε, θα ενισχύσουμε τα κεκτημένα του Σέγγεν και θα προχωρήσουμε στην κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων λιγότερη εθνική κυριαρχία και περισσότερη κοινή υπευθυνότητα θα δώσουν λύσεις στις ελλείψεις που σημειώθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξαντλήσει όλες αυτές τις διαδικασίες στα πλαίσια των μηχανισμών αξιολόγησης Schengen. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι οι εθνικές προσπάθειες και η επανεισαγωγή σύνορων ε, στα εσωτερικά σύνορα είναι τεκμηριωμένες για λόγους εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Η περίοδος πέραν των έξι μηνών ε, φτάνει τώρα, τον Μάρτιο ε, τελειώνει, τον Μάρτιο για τη Γερμανία και αργότερα για τη Μάλτα, τη Σουηδία και την Νορβηγία. Εφόσον λοιπόν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να τις διαδεχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είμαι υπέρ των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Αλλά να περιμένουμε τώρα τις εθνικές αποφάσεις για επανεισαγωγή ελέγχων στα πλαίσια της μεταναστευτικής κρίσης χωρίς να προπαρασκευαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν ανεύθυνο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει αμέσως να αναλάβουμε δράση στην εξωτερική, στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμες ενέργειες πληρέστερες και αποτελεσματικότερες και γι' αυτό θέλουμε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οδηγία ερευνητών και φοιτητών, κάτι το οποίο θα προσελκύσει περισσότερα νέα ταλέντα στην Ευρώπη. Να κλείσω τώρα τα θέματα της μετανάστευσης ε, για το μήνυμα που στέλνουμε ε, με τον εξωτερικό έλεγχο των συνόρων. Μια μεταναστευτική πολιτική ανοιχτή, δεκτική αλλά ελεγχόμενη απαιτεί τον πλήρη σεβασμό των κανόνων Σέγγεν. Για να μπορέσει το δικαίωμα στο άσυλο να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο απαιτούνται εναρμονισμένοι κανόνες εφαρμογής. Θα πρέπει εμείς να συμφωνήσουμε σε θέματα όπως τα κοινωνικά ωφέλη, πρόσβαση στην εργασία και στην εκπαίδευση. Δεν αρκούν όμως οι κοινοί κανόνες. Θα πρέπει να εγγυηθούμε και μια κοινού τύπου εκτέλεση των κανόνων αυτών. Απαιτείται λοιπόν μια σύγκληση σε επίπεδο αποφάσεων και νομολογιών. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε εμείς να εφαρμόσουμε ένα σύστημα παρόμοιο το οποίο χρησιμοποιείται και στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας θα ήθελα όλοι να είναι πιο φιλόδοξοι και βολονταριστές στα πλαίσια μιας πραγματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Να αναφερθώ σε ένα δεύτερο θέμα τώρα, το οποίο σας ενδιαφέρει πολύ και ενδιαφέρει και μας, το κράτος δικαίου. Το Δεκέμβριο του 2014, επί Ιταλικής Προεδρίας, το Συμβούλιο της Ένωσης και τα κράτη-μέλη συνεδρίασαν και υιοθέτησαν κάποια συμπεράσματα στα πλαίσια των οποίων ξεκινούν έναν διάλογο σε αιτήσια βάση για να προασπίσουν το κράτος δικαίου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα αυτά ξεκινώντας ένα πρώτο διάλογο για τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Να θυμίσω ότι στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτος δικαίου αποτελεί το κλειδί πάνω στο οποίο αν θέλετε εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση λοιπόν πρέπει να προωθήσει μια κουλτούρα σεβασμού του κράτους δικαίου στο εσωτερικό της. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία έκρινε απαραίτητο ο διάλογος να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της έλλειψης διακρίσεων και της ισότιμης μεταχείρισης. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία εκφράζει την ευαρεσκιά της γιατί οι ανταλλαγές αυτές απόψεων γίνονται με αντικειμενικό τρόπο. Στα πλαίσια του πρώτου διαλόγου τα κράτη-μέλη παρουσίασαν τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και τις δυσκολίες τους. Η ανταλλαγή απόψεων ήταν καρποφόρα και τα κράτη-μέλη πήραν τον λόγο και μετέφεραν τις απόψεις τους σε σχέση με τις εθνικές τους εμπειρίες. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο προχώρησε σε ανταλλαγή απόψεων για την ανταλλαγή στοιχείων και σεβασμό του κράτους δικαίου στην ψηφιακό κόσμο. Πρέπει να υπάρξει σεβαστό, σεβασμός του κράτους δικαίου και στα πλαίσια των συναλλαγών με ψηφιακό τρόπο. Η Προεδρία προτείνει να εξετάσουμε σε βάθος πολλά θέματα βασικά όπως η ελευθερία έκφρασης, η διακυβέρνηση του διαδικτύου, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία θεωρεί ότι η εκκίνηση του πολιτικού διαλόγου χαιρετίστηκε από το σύνολο των κρατών μελών. Οι ανταλλαγές αυτές επέτρεψαν να εντοπίσουμε καλύτερα τους τομείς τους οποίους απαιτείται και σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο περαιτέρω προσπάθεια. Η συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι το πνευματικό και αφηρημένο. Κάθε παρέμβαση σαν παράδειγμα στον τομέα της ε, δικαστικής εξουσίας, κάθε προσπάθεια φήμωσης των μέσων ενημέρωσης, όλα αυτά είναι εξελίξεις αντίθετες με τα ε, κοινοτικά κεκτημένα. Οι συνθήκες είναι ξεκάθαρες σε σχέση με τους κανόνες της Κοπενχάγης. Είναι καθήκον των ευρωπαϊκών οργάνων να καταγγέλουν με ε, ξεκάθαρο τρόπο και να παίρνουν και μέτρα ε, κύρωσης μερικές φορές αν αυτό χρειάζεται. Το θέμα λοιπόν του κράτους δικαίου είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και εσωτερικά. Σε σχέση με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι που έγιναν πριν λίγες μέρες πριν από το Συμβούλιο, τέθηκαν ορισμένα ερωτηματικά σε σχέση με τον σεβασμό της, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ένα τμήμα της συζήτησης τίθεται σε σχέση με το πώς μπορούμε να σεβαστούμε ακριβώς το δίκαιο και τα δικαιώματα καταπολεμώντας αποτελεσματικά. Τίθεται εδώ το θέμα της καταπολέμησης των κήρυγμάτων μίσους και της ισότητας των φύλων. Ο πολιτικός διάλογος που ξεκίνησε με την Προεδρία μας έθεσε τα θεμέλια για ένα επικοδομητικό διάλογο που ζητά από τα κράτη-μέλη να σεβασμούν το κράτος δικαίου και τα ενθαρρύνει να κάνουν μια αυτοκριτική ανάλυση. Είμαι βέβαιος ότι ο πρώτος διάλογος είναι ένα πρώτο μικρό βήμα. Οι τελευταίες εξελίξεις ορισμένα κράτη-μέλη απαιτούν περαιτέρω σκέψεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο θέμα του σεβασμού του κράτους δικαίου. Δείξατε εσείς τον δρόμο μέσω του ψηφίσματός σας στις 15 Δεκεμβρίου για τα θέματα της Ουγγαρίας και περιμένω με ενδιαφέρον τις συζητήσεις και για την κατάσταση στην Πολωνία. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος σας ε, για την επόμενη ολομέλεια σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με την άδειά σα ε, τώρα έχουν ζητήσει το λόγο 17 συνάδελφοι. Πολλοί εξ αυτών θα ήθελα να ρωτήσουν όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά θα μπορούσαν να ε, ενδιαφέρονται να θέσουν ερωτήσεις και στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους. Ο Ετιάν θα μιλήσει για 7 λεπτά και το ίδιο θα κάνει και ο Φίλιξ. Αν το κάνουμε ε, στα γρήγορα θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Να δώσω πρώτα το, ε, μετά το λόγο για ερωτήσει στον κύριο Άσελμπορ και να απαντήσει και να φύγει. Ε, και οι συνάδελφοι μετά θα μπορούν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Έτσι λοιπόν είσαι ο επόμενο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι τιμή για μένα να σας παρουσιάζω σήμερα τις βασικές γραμμές των εργασιών της ε, Προεδρίας μας ε, σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Δύο γεγονότα σημάδεψαν τις εργασίες μας στη διάρκεια των έξι μηνών της Προεδρίας μας. Ε, η ε, επίθεση που αποφύγαμε στο Παρίσι στο ε, Ταλής τον Αύγουστο και τα πρόσφατα γεγονότα στο Παρίσι ε, στις 13 Νοεμβρίου. Αυτά οδήγησαν σε μια ζητονισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση βέβαια και την αρχή της αναλογικότητας και τα καταφέραμε και αυτό σε μεγάλο βαθμό χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των εξουσιών που έχει ε, ανάληψης πρωτοβουλειών. Στις 15 ε, Ιουλίου του 2015 όταν είχα έρθει εδώ να απευθύνω και πάλι λόγω σε εσάς, είχατε πει ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι σε πολλούς τομείς. Θα πρέπει να ε, οδηγήσουμε την ανανεωμένη εφαρμογή της ε, στρατηγικής ασφαλείας για το 2015-2020. Θα πρέπει να συζητήσουμε δύο νομοθετικά ζητήματα πολύ σημαντικά με το νέο κανονισμό του Europol και την ε, διαπραγμάτευση για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα PNR, για τα στοιχεία των επιβατών, για να μπορέσουμε να έχουμε μία σειρά από μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας Δημοκρατίας επικεντρωνόμενη κυρίως και στην ε, ε, καταπολέμηση των ξένων μαχητών και της ε, παράνομης εμπορίας όρπλων. προχωρήσαμε σε όλα αυτά τα σημεία. Κυρίες και κύριοι, είναι η τιμή μου να μπορώ να σας ανακοινώσω σήμερα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προοδοί στα θέματα αυτά να σταθώ εν συντομία σε κάποια από τα θέματα τα οποία θα ε, αναλύσω στη συνέχεια. Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αυτό αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα της Προεδρίας μας ε, για τους ξένους μαχητές πέραν από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν είναι σε θέση να σταματήσουμε αυτή τη ροή ξέρουμε μεταναστών ε, και προς ε, ε, περιοχές σύραξης, θα πρέπει λοιπόν να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να αναχαιτήσουμε αυτές τις τάσεις και να προσπαθήσουμε να δούμε και τι κίνδυνο αποτελούν αυτοί οι άνθρωποι κατά την επιστροφή τους στην Ευρώπη να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι ε, πηγαίνουν ε, στις χώρες αυτές ε, λόγω ριζοσπαστικοποίησης και θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης, να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που επιστρέφουν, να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα, έρευνες, μέτρα τα οποία θα πρέπει να ελέγχουν πώς επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, να δούμε τι δυνατότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι να διακινούν πυροβόλα όπλα ε, και να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους, καθώς επίσης να βλέπουμε <clears throat> και τι γίνεται με τη στρατολόγηση νέων πιθανών τρομοκρατών. Στις 20 Νοεμβρίου του 2015 η Λουξεμβουριανή Προεδρία διοργάνωσε μια έκτακτη σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για να συζητήσει ακριβώς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εκεί λοιπόν οι Υπουργοί συμφώνησαν να ληφθούν κατεπήγοντα επιχειρησιακά μέτρα για τα θέματα αυτά. Και αυτά τα μέτρα έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπός. Το Συμβούλιο υπενθύμησε ότι πρέπει κατεπηγόντως να ολοκληρωθεί η οδηγία PNR ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 4 ε, Δεκεμβρίου υπήρξε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο για το κείμενο της οδηγίας, το οποίο ψηφίστηκε και στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ στις 10 Δεκεμβρίου και υπήρχε και μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη θετική ψήφο. Αυτό το νέο εργαλείο λοιπόν αυτή τη στιγμή συσταθεί θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε καλύτερα την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα μέσω ενός αποτελεσματικού και ισορροπημένου κειμένου. Οι Υπουργοί δεσμεύτηκαν επίσης μέσω κοινή δήλωση να χρησιμοποιήσουν ε, τη δυνατότητα να συλλέγουν τα δεδομένα στις ενδοκινοτικές πτήσεις και όπως ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνουν υπόψη τους και τα δεδομένα άλλων οικονομικών φορέων. Όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων, η Προεδρία τον Οκτώβριο του 2015 κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα για τους τρόπους καταπολέμησης του φαινομένου. Μεταξύ των μέτρων τα οποία αποφασίστηκαν, η Προεδρία ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 2015 έναν εκτελεστικό κανονισμό για τους κανόνες για τον παροπλισμό αυτών των όπλων. Στις 18 Νοεμβρίου ο εκτελεστικός κανονισμός εγκρίθηκε, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο. Επιπλέον, το Συμβούλιο είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2016 να υποβάλει μια πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα, μια οδηγία η οποία θεωρείται ότι ε, είναι ευσεβής πόθος και θα πρέπει να βελτιωθεί η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης και η Προεδρία ξεκίνησε αμέσως σε επίπεδο Συμβουλίου να ε, συζητά την πρόταση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Και εδώ θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο. Επίσης εδώ να σας πω ότι ε, επικροτώ την πρόσφατη παρουσίαση της Αρμόδιας Επιτροπής ε, για την Οδηγία για τα Πυροβόλα Όπλα και των Εκρηκτικών που θεωρούμε ότι είναι μέτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, και θα είναι συνοδευτικά των εργασιών στο Συμβούλιο. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας επίσης ε, ε, συνοδεύεται και από την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα. Έγιναν αρκετές εργασίες με στόχο να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα προτείνει λοιπόν μέχρι τις αρχές του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα χρησιμοποιώντας ε, όλο ένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στα πλαίσια της πολιτικής για τα ευφυή e σύνορα ζήτησε να γίνει και μία μελέτη ε, στοχευμένη για τον κώδικα σύνορων ε, Σέγγεν και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 7.2. Θα Υπάρχει δυνατότητα να γίνεται συστηματικό έλεγχο τη ταυτότητα ενό ατόμου, των ταξιδιωτικών του εγγράφων, καθώ επίση και κάποια στοιχεία για το κατά πόσον μπορεί κάποιο να αποτελεί απειλή για την εσωτερική ασφάλεια μια χώρα. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μαλλών και Europol, ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε δύο θέματα. Καταρχάς την ανταλλαγή αστυνομικών και δικαστικών πληροφοριών, κυρίως μέσω Ευρωπόλ, και ε, δεύτερον την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω συνεργασίας ε, των υπηρεσιών πληροφοριών. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συστηματική χρήση και στην ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων. Πρόκειται για μέτρα που αφορούν ε, τους ξένους μαχητές ε, που βρίσκονται στο σύστημα της ΕΝΚΕΝ, να υπάρχει διαλειτουργικότητα στις διάφορες βάσεις δεδομένων και επίσης να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις εργασίες της Ευρωπόλ μέσω ε, ενίσχυσης των βάσεων δεδομένων της υπηρεσίας έγιναν σημαντικά μέτρα τους τελευταίους μήνες, κυρίως όσον αφορά την ε, ε, συστηματική χρήση του συστήματος SIS, για παράδειγμα. Επίσης, κατόπιν παρότρινσης της Λουξεμβουριανής Προεδρίας, ε, έγινε και μία ανάλυση της χρήσης των κρατών μελών των διαφόρων μέσων που υπάρχουν διαθέσιμα. Έχει ξεκινήσει η ανάλυση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την ανάλυση για να παρουσιάσει το 2016 συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχύσει ακόμα καλύτερα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπόλ. Όσον αφορά την ανταλλαγή ε, πληροφοριών, η Προεδρία είναι υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών, ε, ε, διατηρώντας βέβαια κατά νου το γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σίγουρα περιορίζεται βάσει των κανόνων που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να είναι διαφορετική από τη μια χώρα στην άλλη. Ε, το αυτό ισχύει και για την πρόσβαση των υπηρεσιών πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων της αστυνομίας και του δικαστικού, ε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανταλλαγή πληροφοριών όταν ε, οι δράσεις ε, των υπηρεσιών πληροφοριών είναι εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν ε, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου μετά την επίθεση του Σεπτεμβρίου του 2011 μέτρα ε, και επομένω μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά. Ε, η συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ορβηγία και την Ελβετία να, ε, και έχει δεσμευτεί να ξεκινήσει μια νέα πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών για να μπορέσουμε να έχουμε πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών που θα είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και πλήρης. Επίσης υπάρχει μια συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον νέο κανονισμό της Europol. Όπως σα είπα τον Ιούλιο, ως στόχο είχαμε η Ευρωπόλ να διαθέτει μια σταθερή νομική βάση που θα σε επιτρέψει να μεγιστοποιήσει τι δυνατότητε τη ε, στην υπηρεσία των κρατών μελών και σεβόμενη την ε, αρχή τη επικουρικότητα και της προστασίας των ενδιαφερομένων και σας, μπορώ να σας πω σήμερα ότι η αποστολή εξετελέστη. Ολοκληρώνοντας, θα αναφερθώ και στην εφαρμογή της στρατηγικής από πλευράς Προεδρίας ε, της ανανεωμένης ε, στρατηγικής για την περίοδο 2015-2020 σε θέματα εσωτερικής ασφαλείας. Σε θέματα εσωτερικής ασφαλείας η Προεδρία μας αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις, κυρίες και κύριοι. Ε, δεν οφείλεται αυτό ε, μόνο στις εργασίες που είχαμε ξεκινήσει, αλλά τελικά καταφέραμε ε, ε, να έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη και στη δέσμευση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ήταν οι δύο σύμμαχοί μας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Οι επιτυχίες αυτές λοιπόν ανήκουν και σε εσά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ καλή συνεργασία το τελευταίο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ετιέν. Ο Φίλιξ, ε, Υπουργός Δικαιοσύνη τώρα. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας και εσάς Πρόεδρε και όλους τους βουλευτές της Επιτροπής σας γιατί υπήρξε μια εξαιρετική μορφή συνεργασίας από πλευρά σας. Ευχαριστώ και τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ. Χωρίς τη δική σας συνεργασία δεν θα είχαμε πετύχει. Να ευχαριστήσω όλους τους συζηγητές, την κυρία Γκρίσμπεκ, Κίνιτσι, Λαουρεστίν και τον Άλμπρεστ που και οι τέσσερις δούλεψαν με εξαιρετικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με μας και μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε συμφωνίες πάνω σε πέντε πολύ σημαντικά θέματα. Τρία είναι δική σας αρμοδιότητα και δύο γιούρι. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το να βρει κανείς μια καλή ισορροπία ήταν ο στόχος. Τελικά επετεύχθη μια συμφωνία υψηλού επίπεδου. Καταλήξαμε σε ένα διακανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι future-proof θα ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών στην ψηφιακή μας κοινωνία με τις ροές των δεδομένων μειώνοντας τους κινδύνους για την ε, προσωπική μας ζωή. Ενθαρρύνουμε και τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα και ενισχύουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο επιτρέποντας την ανάπτυξη μιας ε, δημοκρατίας και στον τομέα του διαδικτύου. Ε, για την οδηγία. Πετύχαμε έναν προσανατολισμό γενικά στο Συμβούλιο Τζάι της 20 Οκτωβρίου και αυτό μας επέτρεψε να διαπραγματευτούμε μια επιτυχή κατάληξη μαζί σας. Θα υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις κατασταλτικές αρχές και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, κάτι το οποίο θα ισχύσει και για τα εθνικά θέματα και για τα διευρωπαϊκά θέματα ή διεθνή θέματα και θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες από ό,τι στο παρελθόν. Τα προβλήματα που είχαμε τα έφεραν στην επικαιρότητα για μια ακόμη φορά και δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό, αυτά που συνέβησαν στο Παρίσι. Πετύχουμε λοιπόν περισσότερα πράγματα από ό,τι σήμερα. Έγιναν και άλλες προσπάθειες από πλευράς των θεσμικών οργάνων και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι στο ύψος των προσδοκιών των πολιτών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα ψηφιακά θέματα σε ποινικό, στον ποινικό τομέα. Νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια σύμφωνη γνώμη και για τις διαδικαστικές εγγυήσεις και για ici d'un progrès très important pour l'espace judiciaire européen. Le rapprochement des droits procéduraux des États membres renforce l'équité όπως επίσης και των διαδικασιών σχετικών με το τεκμήριο αθωότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα γιατί εμείς εργαζόμαστε όλο και περισσότερο για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί η ποιότητα των αποφάσεων αυτών. Οι διαδικασίες που προανέφερα θα βοηθήσουν και χάρη στις προσπάθειες της κυρίας Κινίτσι και της κυρίας Γκρίσμπεκ κάναμε σημαντικά βήματα σε οδηγίες οι οποίες δεν ακούγονται πάρα πολύ σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης αλλά έχουν βασική θα έλεγα βασικό ρόλο να παίξουν στον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης. Ε, στις υπόλοιπες οδηγίες οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται όχι με πολύ γρήγορες ταχύτητες και οι θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν είναι πάρα πολύ κοντινές. Ελπίζω όμως ότι οι διαπραγματεύσεις θα μας επιτρέψουν του χρόνου να καταλήξουμε κάπου. Για τα νέα ψυχοτρόπα. Μένει ακόμα να γίνει πάρα πολλή δουλειά από πλευράς του Συμβουλίου και το συνειδητοποιούμε για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ε, βασικό θέμα. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία έχει προχωρήσει και υπάρχει στήριξη από το Συμβούλιο στα βασικά άρθρα της λειτουργίας της εισαγγελία αυτής, όπως οι αρμοδιότητες, άσκηση αρμοδιοτήτων και διασυνοριακές έρευνες. Οι διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά έχουν ολοκληρωθεί και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ένας ισχυρός Ευρωπαίος εισαγγελέα, μια εισαγγελία ευρωπαϊκή ισχυρή θα υπάρξει, θα δημιουργηθεί σύντομα. Σε σχέση με την εισαγγελία υπάρχει επίσης ε, και ο αγώνας για την καταπολέμηση των μέσων και των ενεργειών εις βάρος των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εδώ έχουμε ε, συζητήσει και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε σχέση με το ΦΠΑ, αν θα συμπεριληφθεί. Λοιπόν, για την ε, αναθεώρηση του ΖΙΣΤ δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Για να ενισχύσουμε πάντως την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις για να δοθούν κάποιες ποινικέ απαντήσεις στην ριζοστοπαστικοποίηση ε, και την βία. Ε, για να αντιμετωπίσουμε επίσης το μεταναστευτικό πρόβλημα και από πλευράς δικαιοσύνης, το Συμβούλιο έχει πάρει σημαντικά μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας και καταπολέμησης της ξενοφοβίας. Σε σχέση με αυτά τα δικαστικά θέματα έχει σημασία η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργαστεί επίσης ε, και με την βιομηχανία του ίντερνετ για να ελεγχθεί ε, η ρητορική του μίσου στο διαδίκτυο που είναι απαράδεκτη. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια στρατηγική έτσι ώστε να φύγουν αυτά τα μηνύματα μίσους από τα κοινωνικά μέσα και να καταπολεμηθούν σε εθνικό επίπεδο στα, στις χώρες που έχουν κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια μέσα για να το πετύχουν. Θα πρέπει λοιπόν να πρικίσουμε την ποινική δικαιοσύνη με τα μέσα τα οποία απαιτούνται. Ξεκινήσαμε συμβούλια στο Συμβούλιο για να καταλήξουμε και σε κάποιες πρώτες συμφωνίες. Οι συζητήσεις μας στο Συμβούλιο σε σχέση με την διατήρηση των στοιχείων των τηλεπικοινωνιών των δεδομένων των τηλεπικοινωνιών ήταν επικοδομητικές. Η απόφαση της 8ης Απριλίου του 2014 δεν απαγορεύει τη συλλογή και τη διατήρηση των δεδομένων, αλλά θέτει συγκεκριμένες και επακριβείς απαιτήσεις σε σχέση με μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα λοιπόν για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για την δική σας προσπάθεια και για την εξωτερική συνεργασία που πετύχαμε σε συνομοθετικό επίπεδο τους τελευταίους έξι μήνες ή καλύτερα των 4,5 μήνες. Νομίζω πως 7 λεπτά ήταν αρκετά καλά. σα αναπτύξατε τα επιτεύγματα της Προεδρίας. Θυμάμαι πως είχατε πει στην αρχή πως θα τελειώσετε με τον κανονισμό των δεδομένων και γελούσα. Γιατί ξέρετε, όλο μιλάμε για διαφάνεια και κάτι τέτοια πράγματα εκεί πέρα. Α, ναι, εσείς γελάσατε, ναι, ναι. τώρα δεν γελάει κανείς πάντως. Και μπράβο σας. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε πολλούς ομιλητές. Όλοι, λοιπόν, θα μιλήσουν. Δύο λεπτά ο καθένας, σας παρακαλώ. Ξεκινάμε την κυρία Χόλμαϊρ. Μόνικα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την Λουξεμβουργιάνη Πρόεδρια, τους τρεις υπουργού που ήρθαν εδώ και μας εξήγησαν το ότι συνέβη όχι μόνο την τελευταία εβδομάδα αλλά τους τελευταίους μήνες. είχαμε νομίζω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Είχα την αίσθηση πως είχαμε εντατική συνεργασία σε θέματα δύσκολα και είμαι και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και εκεί πέρα πραγματικά μας έκανε πολύ καλή εντύπωση η Προεδρία σας. Λοιπόν, τρία, τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα σχετικά αφορά το κλείσιμο των συνόρων. Ακούω πως ε, θα έχει λυθεί μέχρι το Μάρτιο το θέμα των εξωτερικών συνόρων. Το βλέπετε ρεαλιστικό αυτό, γιατί ο Μάρτιος, τι να πω, απέχει τρεις μήνες. Το βλέπετε ρεαλιστικό αυτό και ποιες λύσεις θα βρούμε για το ενδιάμεσο διάστημα όπου έχουμε ανοιχτά σύνορα εκεί που θα έπρεπε να είναι κλειστά και κλειστά εκεί που θα έπρεπε να είναι ανοιχτά για να το πω ευγενικά. Έχουμε δηλαδή κάποια προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα που θα έπρεπε να τα διασφαλίσουμε. Δεύτερον, μιλήσατε για το κήρυγμα μίσους και την στρατολόγηση. Είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο το ότι γίνεται στρατολόγηση μεταξύ των προσφύγων, γιατί είναι απροστάτευτη, αβοήθητη κτλ. Συγκεκριμένα λοιπόν ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο για την στρατολόγηση ειδικά ανασφαλών νέων, ανεξαρτήτως το εάν είναι ήδη στην Ευρώπη ή αν έρχονται τώρα. Και βεβαίως το κήρυγμα του μίσους δεν αντιμετωπίζεται μόνο με διάλογο, αλλά ε, να το πάρουμε σοβαρά. Όταν κάποιος παρακινεί σε δολοφονίες, ε, βίες πράξεις ε, ή ξυλοδαρμό γυναικών ή οτιδήποτε. μιλήσατε για τα δεδομένα. Μιλήσατε για διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων. Είχαμε κάποιους ε, τρομοκράτες που έχουν καταγραφεί τρεις και παρόλα αυτά δεν τους ε, εντόπισαν. Ε, δεν είναι καλό σημάδι αυτό, έτσι. Και για άλλους υπόπτους, αλλά αθώους. Τι κάνουμε για την ε, σύγκριση δεδομένων μεταξύ ΣΥΣ και κρατών μελών σας ευχαριστώ, Birgit Σίπελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν σίγουρη πως πολλοί συνάδελφοι ε, θα έχουν ερωτήσεις, οπότε θα είμαι σύντομη. Για την ζώνη Σέγγεν. Έχω μια ερώτηση γιατί εγώ έχω μπερδευτεί λίγο για την συζήτηση που γίνεται που λένε ότι έρχονται πάρα πολλοί πρόσφυγες. Ο επίσημος αριθμός Frontex είναι πως φέτος έχουμε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με άλλα επίσημα νούμερα, ένα εκατομμύριο από το 1,5 ε, έφτασαν στη Γερμανία. Οπότε, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δέχονται 500.000 πρόσφυγες. πώς είναι υπερβολικό το βάρος για τις υπόλοιπες 27 χώρες. Δεν βγαίνει δηλαδή. Και μια άλλη ερώτηση. Για την καλύτερη συνεργασία υπηρεσιών ασφαλείας. Αυτό είναι απαραίτητο, συμφωνώ. Αλλά μπορείτε να μου απαντήσετε το γιατί η καλύτερη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας και της αστυνομίας. Αλλά ας μιλήσουμε μόνο για αυτές. Γιατί γίνεται ε, όλο και πιο σημαντική. Γιατί με μονομένα κράτη-μέλη και υπηρεσίες ασφαλείας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε την εθνική ασφάλεια λέγοντας πως είναι μόνο ένα ζήτημα μεμονωμένων κρατών μελών. Βλέπουμε πως οι προκλήσεις προέρχονται από όλο τον κόσμο θα έλεγα. Αυτές οι δύο ερωτήσεις έχω λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μείνατε και εντός του χρόνου. Κύριε Κέρκοπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να υποστηρίξω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν για την συνεργασία που είχαμε με την Προεδρία και το επιβεβαιώνω και εγώ με την έκθεσή μου για τα στοιχεία αεροπορικών και ευχαριστώ την Προεδρία και μάλιστα να δούμε τις παρατηρήσεις που έκαναν όταν πρώτο ήρθαν στην Επιτροπή μας πριν ξεκινήσει η Προεδρία για το ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι ε, τους ξαναείδα και βεβαίως είναι πάρα πολλά, αλλά αν δούμε το τι έχει γίνει, οι διασφαλίσεις για τα παιδιά, παραδείγματο χάρη, που κάποιοι, που κάποιους από εμάς μας απασχολούν ιδιαίτερα. Το πώς βλέπουμε την προστασία των δεδομένων. Το είναι βεβαίω, αλλά και το πώς θα πλαισιώσουμε την Europol. Όλα αυτά θετικά πράγματα. Τα μόνο πράγμα στο οποίο μας απογοήτευσαν είναι το θέμα της μεταγκατάστασης και του Δουβλίνου. Έχω τη νέα έκθεση εδώ πέρα για τη μεταγκατάσταση και άκουσα στις παρατηρήσεις πως είχαμε πολύ περισσότερα επιτεύγματα στον ε, τομέα αυτών θεωρείτε πως έχει αλλάξει καθόλου η στάση του Συμβουλίου όσον αφορά την μετεγκατάσταση ή την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Έχει αλλάξει τίποτα. Ε, ελπίζω η Προεδρία να έχει καταφέρει να αλλάξει λίγο την μεταρρυθμιση του δουβλινου εχει αλλαξει τιποτα ελπιζω η προεδρια να εχει καταφερει να αλλαξει λιγο την σταση και την ατμόσφαιρα. Αλλά αυτοί είναι οι τομείς που εμένα με απασχολούν για το επόμενο εξάμεινο και σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ Σόφι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την Προεδρία του Λουξεμβούργου για την καλή δουλειά που έκανε και πράγματι σε πολλές ε, περιπτώσεις που δεν ε, τα καταφέρατε ήταν γιατί έπρεπε βέβαια να συμφωνήσουν και άλλες 27 ε, χώρες. Βεβαίως εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για το πακέτο προστασίας των δεδομένων. Λοιπόν, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Νομίζω πως ήταν μία πάρα πολύ καλή νομίζω αρχή και η Ευρώπη πρέπει βεβαίως να ηγείται δια του παραδείγματος οπότε αν να μιλήσουμε για το πώς θα δείξουμε τις αξίες μας στους ε, νεοαφιχθέντες, ε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε εμείς σε αυτά τα οποία λέμε. Οπότε θα ήθελα να ακούσω λίγα πράγματα παραπάνω, αλλά είμαι και κάπως επιφυλακτική, γιατί κοιτώντα τις κυβέρνηση των κρατών μελών, όλες σχεδόν παραβιάζουν τα δικαιώματα. Ουγγαρία, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Γαλλία, βλέπω μέτρα που λαμβάνονται υπό το κάλυμα της εντρομοκρατίας που δεν έχουν ούτε μία σχέση με το θέμα. Ε, Ρουμανία έχει διαφθορά. Η Δανία, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ψάχνει δια της βίας και θα παίρνει τη μαλφή από τους πρόσφυγες, ε, κάτι το οποίο εγώ βρίσκω ιδιαστικό. Βλέπω δηλώσεις ε, της Βελγίδας ε, Υπουργών Υπουργού Ιστορικών που λέει πως ε, εντάξει το profiling δεν είναι και τόσο άσχημο πράγμα να κρίνουμε κάποιον ανάλογα με την καταγωγή του. Ε, εγώ αυτά βρίσκω ρητορική μίσους ε, από τις κυβερνήσει. Κάθε φορά επίσης μιλάμε για τεράστιες παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Και δεν γίνεται ο κόσμος μας έτσι καλύτερος και ειλικρινά όταν κοιτάω την αντιτρομοκρατία νομίζω πως ε, η ήπειρό μας τα κάνει τελείως λάθος. Γιατί όχι μόνο παραβιάζουμε θεμελιώδη δικαιώματα αλλά είναι και αναποτελεσματική. Αρκεί να δούμε μόνο το τι ακούμε για το πώς αντιμετώπισαν οι βελγικές αρχές ε, την κατάσταση από τις 13 ε, Νοεμβρίου. Μιλάμε για ε, ότι τα θαλάσσουσαν. Οπότε κάθε φορά μας ζητάτε να εγκρίνουμε νέες αρμοδιότητες για τις υπηρεσίες ασφαλείας και επί της δικής σας προεδρίας όταν οι υπηρεσίες σας δεν μπορούν να ξεμπλέξουν τα μπουτια τους. Ε, για ειλικρινά με κουράζει. Και ένα πράγμα θα πω για το PNR. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πρακτικά που θα αναφέρουν τις θέσεις των εθνικών κυβερνήσεων. Νομίζω πως από την απόφαση του ΔΕΚ και πέρα έχουμε δικαίωμα. Γιατί λοιπόν δεν μας λέτε τελικά, δεν, δεν κρατάτε ποια πρακτικά αυτό κάνετε στο Συμβούλιο, οπότε πάλι δεν ξέρουμε το τι γίνεται. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε το τι γίνεται στις συζητήσεις ε, για το PNR με τις θέσεις των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαρζιά. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και τους τρεις ε, για αυτή την ε, γρήγορη περίληψη, η οποία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα προσπαθήσω λίγο τηλεγραφικά να κάνω κάποια σχόλια και ζητώ συγγνώμη διότι συνήθως όταν κάνουμε έτσι λακωνικά σχόλια <clears throat> δεν ε, είμαστε και πολύ διακριτικοί. Έχω αρκετές λοιπόν ερωτήσεις για αυτό το οποίο αποκαλείτε εσείς ε, μεταναστευτική κρίση. Εγώ προτιμώ να την αποκαλώ ανθρωπιστική κρίση και κρίση προσφύγων. Όσον αφορά τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, ε, πολλοί έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, αλλά με ποιον, με την Ερυθρέα, μια χώρα που είναι μια ανοιχτή φυλακή, με το Σουδάν που εξακολουθεί να βομβαρδίζει τον πληθυσμό του, με την Αιθιοπία όπου 75 διαδηλωτές που διαδήλωναν ε, ειρηνικά δολοφονήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Με ποιες συνθήκες συνεργαζόσαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ποιοι είναι οι συνομιλητές σας και πώς διασφαλίζετε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται θα έχουν συνέπειες επιτόπου όπως μας είπατε. Εμένα αυτή είναι η ανησυχία μου. Το γεγονός ότι φεύγει ο πληθυσμός και τη μοίρα του. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος. Ε, στην αρχή μας λέτε <clears throat> ότι ε, θα εγκαταστήσουμε ολικά πάρκα και τώρα ε, φωτοβολταϊκά στην Ερυθρέα. Πραγματικά εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά είναι μέτρα. Όχι γιατί δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφοληθούν από αυτές τις εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ετούντες άσυλο που δεν είναι σε θέση να ζήσουν με αξιοπρεπείς συνθήκες και δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πραγματικά θέλουμε να σεβόμαστε και θέλουμε να δείξουμε ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να δράσουμε. Ε, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι αυτοί που δεν έχουν νομικά δικαιώματα δυστυχώς επαναπροωθούνται. Νομίζω ότι συμπτήσετε λίγο τα πράγματα. <clears throat> Δεν δέχομαι τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού πρόσφυγα. Ε, είναι οι καλοί πρόσφυγες και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θεωρούνται κακοί μετανάστες. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται οικονομική μετανάστευση περισσότερο από ποτέ αρκεί να δει κανείς ε, το παράδειγμα της Γερμανίας ε, για να δει τι δεν κάνουν οι υπόλοιποι. Και ένα τελευταίο θέμα, δυστυχώς εάν βγάλουμε τη Γερμανία από αυτούς που μπαίνουν νομίμως στη χώρα, μειώνεται δραστικά ο αριθμός των ανθρώπων. Επομένως θα πρέπει ε, να ξεκινήσουν νόμιμες οδοί ε, για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν εδώ. Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά την καταπολέμηση της δημοκρατίας και τα διάφορα ζητήματα και το τι κάνουν, δεν θα επανέλθω στο ζήτημα της Δανίας που μόλις ανέφερε πολύ σωστά η Σοφία, αλλά όταν ε, προσπαθούμε να ε, υποχρεώσουμε τους πρόσφυγες που φτάνουν να πληρώνουν ε, τη διαμονή τους και να τους στερούμε τα βασικά τους αντικείμενα, τότε νομίζω ότι κάτι κακό κάνουμε. Όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκου, έγιναν 2.000 έρευνες στη Γαλλία σε δραματικές συνθήκες, ε, ε, υποβάλλοντας τους μουσουλμάνους σε ε, ε, μαρτύρια και από αυτές τις 2.000 έρευνες μόνο δύο άτομα ε, διώχθηκαν και δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Διακόπτει ο Πρόεδρος στην ομιλήτρια. Υπάρχει ένας πολύ μακρύς κατάλογος. Στερείτε χρόνο και από τους συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ λοιπόν προσπαθήστε να μιλάτε για δύο λεπτά γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος. Κάποιοι συνάδελφοι μόλις έχουν ολοκληρώσει τριμερείς διαλόγους και θέλουν να θέσουν ε, συγκεκριμένα ερωτήματα. Προσπαθήστε λοιπόν να περιοριστείτε στα δύο λεπτά γιατί ξέρω ότι μπορείτε να το κάνετε. Ό,τι λέτε μπορείτε να το πείτε και σε δύο λεπτά. Η Τζούντιθ Σαρζεντίνη στη συνέχεια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου πήγε στην Ελλάδα ε, και πήρε προσωπικά θα έλεγα τους 30 πρώτους ανθρώπους που πήγαν στο Λουξεμβούργο. Θυμάμαι τον Επίτροπο Αβραμόπουλο που που βοηθούσε τους ανθρώπους να ανέβουν τη σκάλα, του αεροπλάνο κτλ. Και μετά κοίταξα τα τελευταία νούμερα της ε, τελευταίας επιτροπής. Μετά από αυτού ε, τους 30 δεν υπάρχει τίποτα. Όχι μόνο στο Λουξεμβούργο. Στι περισσότερες χώρες δεν γίνεται τίποτα. Το ερώτημά μου λοιπόν στην Προεδρία του Λουξεμβούργου είναι για εξηγήστε μου εσείς που το παρακολουθείτε. Πώς ε, και δεν ε, μετακινείται κανείς από Ελλάδα και Ιταλία σε άλλες χώρες. Ε, πείτε μας από το Λουξεμβούργο το τι κάνετε, γιατί έχετε 90 θέσεις ε, διαθέσιμες, 90 θέσεις μάλλον καλυμμένες και 520, 520 διαθέσιμες. Και 30 έχετε πάρει μέχρι στιγμής. Δεύτερη και τελευταία ερώτηση. τελειώνει ένα εντατικό εξάμεινο. Αν το Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών ήταν καπνιστής, θα λέγαμε πως με το ένα τσιγάρο άναβε το επόμενο. Και ξέρουμε πως και η Ολλανδική Προεδρία έχει προβλέψει αρκετές συνεδριάσεις. Τώρα λοιπόν μπορείτε να μας πείτε το τι γινόταν στις ε, συζητήσεις. Η κυρία Νετφέλτ ζήτησε πρακτικά. Εγώ θέλω να καταλάβω την ατμόσφαιρα. Γιατί κανείς δεν κοιτάει πλέον την ευρωπαϊκή σκοπιά. Ο καθένας κοιτάει όλον αυτόν τον ωραίο μηχανισμό. Βλέπω εδώ πέρα, έχει ο καθένας λέει τον κατάλογο και σκέφτεται τι θα πάθει η δικιά μου χώρα. Δηλαδή ο κύριος Τούσκ που λέει πως πρέπει να τους κρατούμε για 18 μήνες και κανείς δεν ασκεί κριτική, ε, νομίζω πως ε, και αυτό μας δείχνει το ότι κάπου χάνουμε κάποιες ευρωπαϊκές αξίες και θα αντιλαμβάνομαι πως εσείς οι Λουξεμβούργοι έχετε κάπως μια πιο φιλοευρωπαϊκή αντίληψη. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Άσενμπορν βεβαίως πρέπει να φύγει. Μας το είχε πει. Ένα συντονιστής λοιπόν ακόμα και μετά θα ακούσουμε απαντήσεις. Μάιρ λοιπόν ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Λοιπόν, αυτό το οποίο είδα εγώ σε αυτή την ε, Προεδρία, είδα πως είχαμε πάρα πολλές ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής. Για αποτελέσματα δεν ε, ξέρω. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα της πρώτης ε, συνόδου κορυφής ήταν σχεδόν τα ίδια με αυτά της συνόδου της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει τίποτα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξακολουθούν να λονίζουν ελεύθεροι τρομοκράτες. Μήπω θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβετε τις ευθύνες σας όχι ενώπιον μας, αλλά απέναντι στους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνατε για να σταματήσει αυτή η ροή, ετούν τον άσυλο, αλλά και για να τους προστατεύσετε από την ε, τρομοκρατία. Και το ερώτημά μου, το, εμένα το συμπέρασμα μου το τελευταίο εξάμεινο είναι πως η λύση δεν είναι περισσότερη, αλλά λιγότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Έχω λοιπόν Έγγελ, Κόμες, Φαγιόν, Μπόνι, Ντεπρέ, Στίβενς, Τσιτσόφσκι. Bjork, um, Natalie Griesbeck and Mario I'm going to take all those colleagues. Όλους αυτούς λοιπόν τους συναδέλφους θα τους ακούσουμε μετά από τις ε, απαντήσεις ε, για ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου τον κύριο Άσελμπορν που έχει να πάει στο Συμβούλιο. Ναι, πρέπει να φύγω, να πάω στην Κύπρο. Είναι μία από τις τελευταίες αποστολές ε, που μου ζητήθηκε να κάνω. Μου συστήθηκε μάλλον να κάνω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, αλλά θα απαντήσω γενικότερα στα ερωτήματα τα οποία τέθησαν. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα. Τα εξωτερικά σύνορα, νομίζω εσείς ρωτήσατε κυρία Χολμάιερ, εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι εάν δεν υπάρχουν μέσα το συντομότερο δυνατόν για να ελέγξουμε τα εξωτερικά σύνορα, η Σέγγεν θα καταρρεύσει και κανένας δεν θα μπορέσει να τη διασώσει. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που δεν ελέγχει τα εξωτερικά της σύνορα. Και όταν λέω ελέγχει, δεν λέω τίποτα άλλο, απλώς να ξέρουμε ποιος χτυπάει την πόρτα μας, ποιος θέλει να μπει και ποιος χρειάζεται διεθνή προστασία. Επομένως πρέπει τουλάχιστον να το γνωρίζουμε αυτό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο Είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ε, σίγουρα, αλλά νομίζω ε, δεν είμαι πάρα πολύ αρνητικός ε, μετά από το εξάμεινο και από τα, μετά από τις αρκετές επισκέψεις στην Ελλάδα και τα Συμβούλια Δικαιοσύνης και εσωτερικών Υποθέσεων που ε, διάρκησαν πάρα πολλές ώρες, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι πλέον ε, έτοιμη να δεχτεί τη βοήθεια των ε, οργανώσεων του ΟΗΕ. Δεν είχε τέτοια διάθεση στην αρχή και των ευρωπαϊκών οργανισμών. νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου που είναι αρκετά αμφίσιμες αλλά αν ε, ε, μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε θα μπορέσουμε ίσως να καταλήξουμε κάπου. Υπάρχει μια μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρότεινε ακτοφυλακές καθώς επίσης και πήγιους και χερσαίους ελέγχους, ε, να υπάρχει ακτοφυλακή και στη θάλασσα και στην ξηρά. Επομένως, ο έλεγχος των συνόρων δεν είναι υπόθεση μόνο των χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είναι ένας ρόλος ο οποίος θα πρέπει να ε, αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση. Και πραγματικά εγώ φρονώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις ταχύτατα. Όσον αφορά το θέμα των αριθμητικών στοιχείων. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε εμείς είναι ότι φέτος είχαμε 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους που διέσχισαν τα ευρωπαϊκά σύνορα. 1,5 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο 60.000 ζήτησαν διεθνή προστασία. Νομίζω ότι η κυρία που έθεσε την ερώτηση έφυγε, αλλά αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε. Τώρα, όσον αφορά την μετεγκατάσταση και την ε, επανεκατάσταση. Από την πρώτη συζήτηση που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολύ πιο εύκολο να βρούμε μια λύση για την ε, επανεγκατάσταση από ότι μια λύση για τη μετεγκατάσταση. Ξέρετε τη διαφορά. Ε, relocation, επανεγκατάσταση, είναι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απλώς θα τους πάμε αλλού ε, και μετεγκατάσταση είναι όταν τους έχουμε στην Τουρκία, στην Ιορδανία ή οπουδήποτε αλλού και θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο. Υπήρχε μια χώρα που είπα αμέσω ότι δεν έχουμε ε, επανεγκατάσταση και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μόνο μετεγκατάσταση. Σε γενικές γραμμές δεν θα λειτουργήσει κατά την άποψή μου η επανεγκατάσταση στους τρεις-τέσσερις πρώτους μήνες. Και δεν φταίει η Ελλάδα, δεν φταίει η Ιταλία, φταίει το σύστημα το οποίο ακόμα δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Η Ελλάδα κάνει πολλές προσπάθειες ε, στα πέντε μεγάλα νησιά και νομίζω τους τελευταίους μήνες τα πέντε μεγάλα νησιά τα οποία βρίσκονται ε, κοντά στις ακτές της Τουρκίας είχαν hot spot που ήταν αποτελεσματικά. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν διάφορα σκάφη στα νησιά και φτάνουν μετά στον Πειραιά, ε, εκεί έγινε το πρόβλημα γιατί αυτοί μετακινούνται προς το βορρά. Η Ελλάδα είπε ότι είναι διατεθειμένη να έχει πολύ μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής ε, στην ενδοχώρα. Το ιδανικό θα ήταν με βάση αυτό να συζητήσουμε με τους ε, ε, μετανάστες και να οργανώσουμε τη μετεγκατάστασή τους σε συνεργασία με το Frontex και την Υπηρεσία ασύλου και ούτω καθεξής. Είπα ευθύ εξ αρχής ότι δεν πρέπει να καταστρέψουμε τους διάφορους μηχανισμούς γιατί θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν το, στο μέλλον. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η κρίση δεν θα διαρκέσει ένα, δύο, τρία χρόνια, μπορεί να διαρκέσει και μια δεκαετία, επομένως θα χρειαστούμε ένα συστηματικό τρόπο να ε, επαναπροωθούμε τους ε, μετανάστες που έρχονται να χτυπήσουν την πόρτα μας. Η προσωπική μου εντύπωση μετά από το τελευταίο συμβούλιο Τζάι ήταν ότι αν γνωρίζουμε ευθύ εξ αρχής ότι τώρα δεν λειτουργεί το σύστημα, ίσως θα έπρεπε Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Σύριοι οι οποίοι χρειάζονται διεθνή προστασία στην Τουρκία, μήπως θα έπρεπε να πάμε στην Τουρκία και να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 50.000 ανθρώπους και να τους εφα... Ε, ε, ε, αφαιρέσουμε από το ποσό της μετεγκατάστασης. Έτσι θα μπορέσουμε να πούμε ότι θα ξεκινήσει μια πρώτη λύση. Και να μην μιλάμε μόνο με οικονομικά μέσα ή με θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων, αλλά να είμαστε και διατεθειμένοι να δεχτούμε και μια επιβάρηση. Αυτή είναι μια ιδέα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στους επόμενους ε, μήνες, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις για τη μετεγκατάσταση. Σας είπα την άποψή μου. Το σύστημα δεν θα πρέπει να καταστραφεί. Κατά την άποψή μου θα μας χρησιμεύσει στο μέλλον, αλλά προς το παρόν δεν είναι ο μηχανισμός που χρειαζόμαστε προκειμένου να κάνουμε ανακατανομή των φαρών και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευφυείς, και ίσως με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε ίση κατανομή καθηκόντων και να μην ε, ε, έχουμε τόσα προβλήματα οργανωτικά. Όσον αφορά το κράτος δικαίου τώρα, κυρία μου αναφερθήκατε στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στη Δανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να σέβεται όλα όσα και εσείς και εγώ ε, πιστεύουμε ότι ισχύουν για το κράτος δικαίου και βλέπουμε στι διατάξει του κράτους δικαίου. Εγώ δεν είμαι σε θέση να πω σε μια χώρα όπω η Γαλλία που αντιμετωπίζει όλα όσα αντιμετώπισε και με όσα συνέβησαν στις 13 Νοεμβρίου να του πούμε ότι ό,τι κάνετε είναι παράλογο. Ε, Ξέρω ότι είστε ευρωβουλευτή, ε, δεν το φαντάζομαι, είστε ευρωβουλευτέ, έχετε δικαίωμα να εκφράσετε την άποψή σα, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή, αν γίνει η συζήτηση στο Συμβούλιο για το κράτος δικαίου, είναι να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις ε, από τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης λένε ότι το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την κάνουν να διαφέρει ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφερειακές οργανώσεις είναι ότι οι αξίες αυτές πρέπει να γίνονται σεβαστές. Και βλέπουμε σε μια χώρα όπου ξαφνικά μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση η δικαιοσύνη να μην είναι αυτή που πρέπει να είναι, να υπάρχουν παρισφρήσεις και δεν είναι πλέον αυτόνομη και ελεύθερη η δικαιοσύνη και πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Το είδαμε σε κάποιες χώρες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι υπάρχουν τρόποι να δραστηριοποιηθούμε ε, ώστε να μην είναι απόλυτα ελεύθερα τα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να τα αναλύσουμε πάρα πολύ καλά, να επικρίνουμε και εάν χρειάζεται να διαβάσουμε και τις συνθήκες και να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Από πολιτική σκοπιά πρώτα βέβαια, αυτό είναι σαφές, και πρέπει όμως να καταφέρουμε να βρούμε και λύσεις οι οποίες θα είναι γραμμένες στις συνθήκες και να είμαστε και λίγο πιο σαφείς. Τώρα, αν θα γίνει στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σημασία. Διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες πραγματικά πηγαίνουν προς κατευθύνσεις που δεν είναι αντάξιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του πώς αντιλαμβάνεται τις ε, βασικές θεμελιώδεις αρχές. Η συζήτηση που έγινε τον Νοέμβριο ήταν μια ακαδημαϊκή συζήτηση σε μια ωραία αίθουσα ε, πραγματικά την επόμενη φορά πιστεύω ε, βέβαια ότι αυτό θα είναι ε, ήδη επί Ολλανδικής Προεδρίας θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σαφείς και ξεκάθαροι και πραγματικά εάν ε, πρέπει να τιμωρήσουμε μια εξέλιξη σε μια χώρα που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίζει να κινηθεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι πρεσβεύουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το κάνουμε και εκεί θα πρέπει να ε, δημιουργηθούν και κάποια ερωτηματικά, να δούμε κατά πόσο βρισκόμαστε πια σε ένα σύστημα το οποίο ε, είναι αντίστοιχο του Σοβιέτ, της Σοβιετικής Ένωσης. Σε κάποιες ερωτήσεις ε, τέθηκε και το θέμα των αιτίων, τα βαθύτερα αίτια της ε, μετανάστασης. Πολύ σωστά κυρία Βερζιά αναφερθήκατε στην κατάσταση στην Ερυθρία και το τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι πολύ σωστό να ξαναστείλουμε τους ανθρώπους εκεί. Στην Ερυθρέα ε, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν, από την Ερυθρέα δεν ε, τους στέλνει ξανά κανείς αυτή τη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να ε, βρούμε λύσεις για την πηγή αυτών των μεταναστευτικών ε, ροών. Έχουμε ίσως κάποιες ελπίδες στη Λιβύη. Είμαι υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και ο κύριος Κόμπλερ, ο οποίος είναι ένας Γερμανός διπλωμάτης που ανέλαβε ε, μετά από τον Περναντίνο Λεόν και μετέβη στην Τρίπολη και έχουμε κάποιες εξελίξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά η μόνη δυνατότητα να εμπλακούμε ως Ευρωπαίοι και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρούμε ένα πεδίο συνεννόησης με τις λιβικές αρχές είναι αυτή. Θα ήταν πάρα πολύ θετικό και ε, όσον αφορά τη συνεργασία μας, αλλά και όσον αφορά μια πιο λογική αντιμετώπιση των μεταναστών που έρχονται από εκεί. Ε, ξέρετε επίσης ότι ε, έγιναν κάποιες συνεδριάσεις ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε ελπίδες και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να σταματήσει αυτή η σφαγή στη Συρία. Δεν μπορούμε διπλωματικά να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Ισλαμικό κράτος, με τους βαρβάρους, αλλά νομίζω ότι το μήνυμα ελήφθη και νομίζω ότι αυτή ε, η νέα συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους αν δείτε και τους δύο ε, επικεφαλείς, τον Κέρι και τον Λαυρόφ, ε, ίσως μπορούν να μας δώσουν κάποιες ελπίδες. Και αν τελικά τα καταφέρουμε στη Συρία, θα μπορέσουμε ίσως να τα καταφέρουμε να έχουμε και μεγαλύτερη σταθερότητα στο Ιράκ. Το μόνο, το άλλο σημείο κλειδί είναι η Τουρκία. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τουρκία σε πολλά θέματα. η διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας με τους Κούρδους και η ε, επιδίωξη στρατιωτικών λύσεων. Πρέπει να δούμε όμως ότι η Τουρκία έχει υποδεχθεί μέχρι τώρα 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία. Ξέρω ότι το θέμα αυτό προκαλεί συζητήσεις αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία δις προς την Τουρκία δεν είναι μια βοήθεια προς την τουρκική κυβέρνηση, αλλά είναι μια βοήθεια έτσι ώστε τα παιδιά των οικογενειών από τη Συρία να πάνε σχολείο, να υπάρχει ιατρική φροντίδα και οι γονείς των παιδιών αυτών να έχουν την προοπτική να βρουν μια θέση απασχόληση στην Τουρκία. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε φυσικά τις αιτίες της σύγκρουσης και αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θα πρέπει να δώσουμε έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την πολεμική σύγκρουση. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο των άλλων, πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο γιατί όπως σας είπα θα επισκεφθώ την Κύπρο και τη μία πλευρά και την άλλη, την επίσημη πλευρά λέει ο μιλητής από τη μία αλλά και τους άλλους από την άλλη. Um, ευχαριστώ, Ετιέν. Έχει αλλάξει λίγο η ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Τα έχω μπλέξει. Θέλω να πω ευχαριστώ Ζαν και όχι ευχαριστώ Ετιέν. Έχω μια μικρή σύγχυση λέει ο κύριος Μωράς. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι ζητώ συγγνώμη αν είχατε συγκεκριμένε ερωτήσεις για τον Υπουργό Άσεμπορν. Οι συνάδελφοι θα προσπαθήσουν να δώσουν τις απαντήσεις που θέλετε. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών. Ο επόμενος. Ο κύριος Σέγγελ, ο οποίος ομιλεί την Λουξεβουργιανή διάλεκτο. Λοιπόν, ε, συγχαρτία για την επιτυχημένη Προεδρία. Αυτά, είναι, αυτά που είπα Κλώδη ήταν σε μια γλώσσα που υπάρχει αλλά δεν είναι επίσημη βεβαίως. Λοιπόν, Ζαν, θετικό το ότι πας στην Κύπρο, καλή ιδέα, γιατί εγώ ε, Βεβαίω επέμεινε να το κάνεις πριν τελειώσει η Προεδρία και πες στους Τούρκους ότι με το να μειώσουν κατά 3 δισεκατομμύρια το κόστος κατοχής στη Βόρεια Κύπρο δεν θα χρειαζόταν το 3 δις που τους δίνουμε εμείς για τους πρόσφυγες που πάνε ούτως ή άλλως στα σύνορά τους και έχουν ε, υποχρέωση να τους περιθάλψουν όπως και εμείς. Έχω ε, υπάρχει, πρόβλημα κράτους δικαίου με αυτή τη χώρα. Δεν είμαι αντιτούρκος, έτσι, ποτέ δεν ήμουν. Αλλά έχουμε ένα πρόεδρο που δεν εμφανίζεται καν. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός εμφανίζεται και μετά βγαίνει στις κάμερες και λέει «Μια χαρά, θα ανοίξουμε νέα κεφάλαια, θα πάρουμε τρία δις». Αρκετοί θα μπαίνουν χωρίς βίζα κτλ. Αυτό θα ήταν διανόητο πριν από έξι μήνες για σωστούς λόγους. Και αφού το δεχτήκαμε αυτό, αρχίζουν πάλι να βομβαρδίζουν τον ίδιο τους το λαό. Ε, ε, λίγο περίεργα όλα αυτά. Και ίσως μας τη φέρανε, μας πιάσανε κότσους που λέμε. Και ε, από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο πρόεδρος. Ε, λέει ο Ζαν θέλει να απαντήσει πριν φύγει. Απλά για να πω το μήνυμά σου για εμένα. Ε, πήγες εσύ στην Κύπρο, προσπάθησε να είσαι και επικοδομητικός, εγώ θα το κάνω, θα έχω το μήνυμά σου κατά νου, αλλά για να είμαστε πραγματικά επικοδομητικοί για μια λύση η οποία ίσως να μην απέχει πολύ νομίζω πως δεν χρειάζονται λόγια τέτοια επιθετικά εγώ δεν είμαι βουλευτής αυτή τη στιγμή αλλά τα λόγια αυτά δεν θα βοηθήσουν πρέπει να είμαστε έξυπνοι αλλά να στείλουμε το μήνυμα που σωστά ε, ήθελες να μεταφέρω στην Κύπρο. Αυτά. Did you want to conclude, Frank? Just... Frank, ναι. Ολοκλήρωσε. Μα το, το μήνυμα αυτό ήταν για την ε, τουρκική δημοκρατία, έτσι. Ούτε καν για τους τουρκοκύπριους να ολοκληρώσω για το κράτος δικαίου. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες μιας διαρθρωτικής καταπάτησης του κράτους δικαίου για διάφορους λόγους, είτε για διολογικούς λόγους στην Ουγγαρία, στην Πολωνία ή και κάπου αλλού, με πρόσφυγμα τις ε, ε, προκλήσεις για την ασφάλεια όπως στη Γαλλία ή όπως και αλλού, αλλά πραγματικά είμαστε μάρτυρες γεγονότων που με φοβίζουν. Ε, αναφέρθηκε σε μια σοβιετική εντύπωση σε σχέση με την Πολωνία. Εγώ έχω μια τελείως χειρότερη άποψη. Αν πρέπει να δεχτούμε επαόριστον, για παράδειγμα, να γίνονται έρευνες 24 ώρες 24 ώρο, να μπαίνουμε σε σπίτια ανθρώπων μέσα στη νύχτα, χωρίς ε, έγκριση ανακριτή ε, και να μην ε, απελευθερώνονται αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω ότι αυτή είναι παραβίαση μακροχρόνια και νομίζω ότι ουσιαστικά είναι ακραίες λύσεις για την αντιμετώπιση των φόβων που έχουμε για την τρομοκρατία, διότι θα αποσταθεραπήσουμε τον κόσμο και δεν θα προσφέρουμε καμία ασφάλεια. Ευχαριστώ. Λιάννα Γκόμες. Κρίμα που φεύγει ο κύριος Υπουργός. Τέλος πάντων έχει και δουλειές βέβαια. Έχει να πάει και στην Κύπρο. Και ελπίζω να φτάσει το μήνυμα και στην Τουρκία. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση ήταν για τον κύριο Άσελμπορν, αλλά τελικά θα απευθυνθώ στους άλλους υπουργούς, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνανε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. συζητάτε για οικονομικές ε, κυρώσεις ε, απέναντι στις χώρες που δεν ε, τηρούν τα της επαναγκατάστασης. Δεν ξεχνάω βεβαίως τα όσα ζητήσαμε για την Ουγγαρία. Αλλά ακριβώ επειδή υπάρχουν και άλλες χώρες, ανέφερε την Πολωνία ο κ. μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Σκέφτεστε μήπως οι οικονομικέ κυρώσει. γιατί χώρες σαν τη δικιά μου την Πορτογαλία που θέλει να πάρει περισσότερες πρόσφυγες θα έπρεπε να υποστηρίζονται, ενώ όσοι δεν είναι διατεθειμένοι θα έπρεπε να τιμωρούνται για την έλλειψη αλληλεγγύης. Μίλησε ο υπουργό για την ανάγκη να δούμε το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Μα τι έχει κάνει το Συμβούλιο για να ανοίξει νόμιμες διόδους. Μήπως αυτό θα ήταν ο έξυπνος τρόπος για να υπάρχει έλεγχος των συνόρων. Γιατί ο έλεγχος των συνόρων, ας είμαστε ειλικρινείς, Δεν γίνεται έτσι διάταγμα και να γίνει δεν θα εφαρμοστεί όπως ξέρουμε. Και βεβαίως όπως είπαν και άλλοι δεν γίνεται να επιστρέφουμε κόσμο στην Ερυθρέα και στην Αιθιοπία. Κάτι άλλο. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Και για το ότι δεν ε, είναι υποχρεωτικό αυτό μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Γιατί. Δεν κάνουμε αυτό που έγινε στην Europol. Να δούμε εάν γίνεται κοινή χρήση των εθνικών βάσεων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, γιατί μάλλον δεν γίνεται. Και τέλος το παραθυράκι. Αν θέμε να ελέγχουμε τα σύνορα, γιατί το παραθυράκι των ιδιωτικών αεροπλάνων στα PNR γιατί οι περισσότεροι έμποροι όπλων το παίζουν businessmen. Ευχαριστώ, Μπόνι. Ευχαριστώ, θα μιλήσω πανικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λουξεμβουργιανή Προεδρία για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν τους τελευταίους μήνες. Κάποιες βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις έγιναν ήδη δεκτές. Να κάνω όμως τρία σχόλια. Πρώτον, για την αλληλεγγύη και την προστασία των συνόρων. και τη στάση μας απέναντι στους πρόσφυγες. Νομίζω ότι καλό θα ήταν για όλους να αντιμετωπίσουμε αυτό το άγχος το οποίο μας έχει πιάσει όλους. Ένα άγχος που τροφοδοτείται από μια στάση εναντίον των προσφύγων και τον μύθο που καλλιεργείται επί τη βάση του άγχους αυτού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα καταρχάς ε, της ρητορική μίσους. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την τρομοκρατία, αυτό αφορά και αυτόν τον νεοεθνικισμό ο οποίος έχει αρχίσει να αναδύεται σε διάφορες χώρες. Αυτή η ρητορική του μίσους δυστυχώς επιτρέπει να δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι τους οποίους σιγά σιγά καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Τώρα για τα ψυχοτρόπα. Εγώ συμμερίζομαι με τις ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν από την Προεδρία και για την κατάσταση στην δική μου χώρα, όχι μόνο σαν μέλος κόμματος αλλά σαν Πολωνός πολίτης μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει σε σχέση με αυτό συλλήψεις. Ο κ. Ντυπρέ. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία με κάθε ειλικρίνεια και για τα θέματα που μας αφορούν και για τα θέματα της Επιτροπής Προϋπολογισμών έκανε εξαιρετική δουλειά και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Να σχολιάσω λίγο προς τη Σοφή γιατί σε σχέση με τη δική μου χώρα στάθηκε λίγο υπερβολική. Νομίζω ότι οι χώρες οι οποίες δεν γνώρισαν θύματα, θα έλεγα 130 άνθρωποι που τους φάξανε σαν τα μαύρα σκυλιά στο δρόμο, νομίζω ότι δημιουργούνται ευαισθησίες και αντιδράσεις διαφορετικές από αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα σε εισαγωγικά την έχουν βγάλει καθαρή. Λοιπόν, είπατε ότι και το είπε η Σοφή και δεν διαφωνώ μαζί της, ε, θα κατάσχονται τα προσωπικά αντικείμενα και τα τιμαλφή των προσφύγων για να πληρωθεί το κόστος της ε, διατήρησής τους, συντήρησής τους, φροντίδας τους κτλ. Ποια είναι η άποψή μας, μπορείτε να αφήσετε ασχολία στο μια τόσο ηλίθια φράξη. Τώρα πάνω από ένα εκατομμύριο αυτό θα κοστίσει φυσικά, θα χρηματοδοτήσουμε τα hot spot αλλά κυρίως ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να βρουν δουλειά, να ενσωματωθούν κτλ. Μήπως ε, τα ταμεία συνοχής εδώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ε, των προσφύγων εν μέρη. Έχουμε και στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών την αλλαγή των κριτηρίων χρήσης των ταμείων αυτών. Τώρα, για του συστηματικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, για τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κοιτάξτε, αλλά δεν τροφοδοτούμε το σύστημα Σέγγεν. 14 χώρες δίνουν στοιχεία στο Σέγγεν και δεν είναι καν υποχρεωτικό. Δεν έχουμε, θα έλεγα, ξεκάθαρους ορισμούς για θέματα μικροτρομοκρατίας, για θέματα ε, ορισμού του τι είναι ένας ξένος μαχητής λοιπά. Πολλές ερωτήσεις αλλά δεν έχω χρόνο άλλο. Κινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και τους παρόντες υπουργούς για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον κύριο Μπράζ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε σε ένα πλαίσιο πραγματικής συνεργασίας για τις διαδικασίες ε, για τους ανηλίκους που εμπλέκονται σε ποινικέ δικαστικές έρευνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά ήταν πολύ περίπλοκη η οδηγία. Τον ευχαριστώ για την τεράστια προσπάθεια που έγινε ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποιους σωστούς στόχους. Έτσι πιστεύω ότι έχουμε πετύχει. Είναι η πρώτη οδηγία στον τομέα αυτό, στον κλάδο αυτό αν θέλετε και πρόκειται για ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο το οποίο επιτρέπει και την κατανομή των ποινικών ευθυνών όπως επίσης και λαμβάνει συνεχώς υπόψη το εύθραυστο, το ευάλωτο της συγκεκριμένης ηλικία. Είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να χαρακτηρίζει το σύνολο του χώρου δικαστικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ λοιπόν την τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε στο συγκεκριμένο τομέα το Συμβούλιο. Τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις έτσι κι αλλιώς και σε τομείς οι οποίοι με ενδιαφέρουν και εμένα. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που ακούστηκαν αλλά θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς τους δύο υπουργούς. Το θέμα της μετανάστευσης θέτει ένα άλλο θέμα το οποίο εφήγεια θα έλεγα επιδερμικά το θέμα της καταπολέμησης ε, των σωματεμπόρων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ε, είναι στην επικαιρότητα στα πλαίσια της, της τραγωδίας αυτής της νέας μορφής μετανάστευσης. Πρόκειται για μια εγκληματική θα έλεγα δραστηριότητα που συνδέεται και με θέματα διαφθοράς, παρανομοχρηματοδοτήσεων χρηματοδοτήσεων κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το σχολιάσετε και να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και ποιος είναι ο χρονισμός έτσι ώστε στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να ακουστεί και να συνεισφέρει στην καταπολέμηση αυτού του τύπου της εγκληματικότητας. Η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους να ευχαριστήσω και εγώ τη Λουξεμβουριανή Προεδρία για την εξαιρετική της δουλειά. πάνω στα θέματα που ασχολήθηκε η Επιτροπή μας. Και όπως είπε και η Κατερίνα, στο θέμα ακριβώς που προανέφερα προηγουμένως, το euh, τεκμήριο της αθωότητας. Η Προεδρία είναι όμως ο διευθυντής της ορχήστρας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει και να διορθώσω δεν μιλάμε για τη Βαλερή Τριβάιλερ αλλά για την Κατρίν Τριβάιλερ και αυτό έχει σημασία. Το λέω αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά πραγματικά η Προεδρία ήταν πολύ αποτελεσματική γύρω από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε. Τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις ή σχόλια καλύτερα. Έχουν τεθεί πάρα πολλές ερωτήσεις και δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Τρία όμως η μία επανέρχεται η κυρία Γκρισμπέκ. Θα συμφωνήσω εδώ με την Καταρίνα. Δεν είχαμε κάνει ένα πακέτο για την βοήθεια τη διαδικαστική και τα δικαιώματα τα διαδικαστικά για τα παιδιά και το τεκμήριο αθότητας. Δεν κάναμε ένα πακέτο σε σχέση με αυτό. Αλλά όμως υπογραμμίσαμε την ανάγκη να κινηθεί το Συμβούλιο για το τρίτο σκέλος αυτού του μη πακέτου που αφορά την έκθεση De Jong για την διαδικαστική βοήθεια. Υπάρχουν οικονομικές πλευρές, υπάρχουν διαδικαστικές πλευρές, διάφορες χώρες κολλησιεργούν, κάνουν ότι δεν ακούν, αλλά νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να υπάρξει μια κάποια εναρμόνιση και αποτελεσματικότητα στα αρχικά κείμενα. Το δεύτερο σημείο, πάρα πολύ σύντομα, δεν είμαι πρωτότυπη σε σχέση με αυτό. Μου φαίνεται ότι θα ήταν σωστό και συμφωνούν πολλοί συνάδελφοι να προχωρήσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. και όχι να έχουμε αυτό το αίσθημα που νιώθουμε τώρα ότι στην ουσία πηγαίνουμε ανάποδα σε, ένα, σε μια ηλεκτρική σκάλα. Ε, και ένα τρίτο σημείο το οποίο δεν έχει τεθεί μέχρι τώρα νομίζω και είναι μια παρατήρηση, ερώτηση θα έλεγα για το τι θα ακολουθήσει στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας υπάρχει το θέμα της, ε, κατα, ε, της διαγραφής της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Ε, φυσικά εδώ συνεργαζόμαστε με τα διάφορα δίκτυα και με τις διάφορες επιχειρήσεις τις διαδικτυακές, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρξει μια πιο ενιαία αντίδραση από πλευράς των κρατών μελών γιατί ορισμένες χώρες από τις 28 δίδουν κάποια χρήματα για να ελέγχεται το διαδίκτυο, άλλες χώρες όμως δεν το κάνουν αυτό και η Ευρώπη εδώ μάλλον θα πρέπει ε, να προσφέρει κάτι περισσότερο. Και θα κλείσω τώρα ε, λέγοντας ότι σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο και με το περιεχόμενο ρητορικής μίσους δεν έχουμε κάποιους ορισμούς κοινού. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός για τα όρια των ενιών αυτών. Ίσως λοιπόν για να είμαστε πραγματιστές και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε να βρούμε κάποια λύση. Thank you. Next is Thomas please. Συνέχεια ο κύριος Σντόσκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Εγώ βέβαια συνήθως ακούω ότι μου λένε θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλήσω εντός των χρονικών ορίων. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτούς που ε, εγκομίασαν το έργο της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Ε, κάνατε εξαιρετική δουλειά το, στη διάρκεια του εξαμήνου και σας ευχαριστώ γι' αυτό διότι μετά την Ιταλική Προεδρία θα θεωρήσω ότι είστε η υποδειγματική Προεδρία. Ό,τι είπατε το κάνατε. Τώρα, για τα hot spots, ε, συμφωνώ απόλυτα, έγιναν πολλά πράγματα από πλευρά Ελλάδος, αλλά πώς εξηγείτε το εξή. Εγώ το τελευταίο το περασμένο Σαββατοκύριακο ήμουνα στα σύνορα ε, με την Φύρομ και από την Αθήνα κυκλοφορούν κανονικά ε, λοφορεία πούλμαν με 50 ευρώ χρέωση και επομένω φτάνουν μέχρι τα σύνορα. <clears throat> Πολύ συχνά πρόκειται και για οικονομικούς μετανάστες. Αυτή δεν είναι όλη αυτή η παράλογη κατάσταση των κρατών. Στην πραγματικότητα δηλαδή νόμιμα μεταφέρονται άτομα από, τη μία χώρα, από το ένα σημείο στο άλλο. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια μπίζνα. Πρόκειται για τη χειρότερη επιχείρηση. Αφορά ανθρώπους, ταλέπορους που ε, τους εκβιάζουν για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Europol. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στην Europol εδώ. Η Europol στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα μας είπε ότι όσον αφορά τη διακίνηση ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται και για την διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και το καθεξής. Δηλαδή δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, ε, δίμευσης από νομικής Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να ασχοληθούμε και με αυτά και όσον αφορά τη βάση δεδομένων, αναφερθήκαμε στους ξένους μαχητές. Στη βάση δεδομένων αυτή τη στιγμή της Ευρωπόλη υπάρχουν 17 άτομα, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαβάζει καμία πληροφορία για τους ξένους μαχητές της που πηγαίνουν να πολεμήσουν στη Συρία. Και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι λειτουργικές αυτές οι βάσεις δεδομένων. Αυτή είναι η τελευταία μου και συγγνώμη αν ξεπέρασα το όριο. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Βαν Κάουφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένου του χρόνου θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα μόνο ζήτημα. Και βέβαιως να ευχαριστήσω και εγώ τους τρεις υπουργούς και την Προεδρία για την καλή δουλειά που έκαναν και εύχομαι την αποκαλή ξεκούραση τις γιορτές. Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και Υπουργέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάτε πως ε, θέλετε να ολοκληρώσετε σύντομα τώρα. Το τι σημαίνει σύντομα θα το δούμε. Αλλά γνωρίζετε πως ε, το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα στην απόφαση. Και ε, δεδομένη της προόδου, καλό είναι να ενημερώνετε και το Κοινοβούλιο κάποτε. Παράκλησή μου λοιπόν είναι να μας ενημερώσετε για το τι γίνεται και παρακαλώ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας αν υπάρξει πρόοδος ε, το μότρο δυνατόν να μιλήσουμε με την Ολλανδική Προεδρία του χρόνου για να ενημερωθούμε. Να δούμε δηλαδή ποια κράτη στηρίζουν ή όχι, γιατί εμείς το θέλουμε βέβαια, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και το τι περιέχεται στην πρόταση αυτή αυτά και καλές γιορτές, καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εμεί το θέσαμε το θέμα με την Προεδρία, την ερχόμενη. Με το πρέσβη, το είπα και στην Σίλβια Και ούτως ή άλλως θα έρθει η Προεδρία 11 Ιανουαρίου στην Επιτροπή. Οπότε οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κύριος ε, Χαλα Άχο. Υπάρχει μια νέα οδηγία για πυροβόλα όπλα που αναφέρατε κύριε Σνάιντερ. Συμφωνώ με την Κομισιόν πως καλό είναι να υπάρχουν κάποιες κοινέ προδιαγραφές ε, και κοινού ορισμούς για τα βασικά συστατικά μέρη, να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες κτλ. Όμως υπάρχουν και κάποια στοιχεία ανησυχητικά, συγκεκριμένα η πρόταση απαγόρευσης και κατάσχεσης των ημιαυτόματων νόμιμων πυροβόλων όπλων που ομοιάζουν πολύ με τα αυτόματα. Πώς αυξάνεται έτσι η ασφάλεια. Όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στις πρόσφατες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις και σπανίως χρησιμοποιούνται. Πρώτος πρόταση αυτή δεν θα επηρεάσει ούτως ή άλλως ε, την τρομοκρατία ή το έγκλημα και στην πράξη είναι δύσκολο να απαγορεύσει κανείς κάτι επειδή μοιάζει με κάτι άλλο. Γιατί είναι θέμα μετά εμπειρίας, να μην πω γούστου το εάν μοιάζει ένα ημιαυτόματο με αυτόματο. Και ε, ε, η νομοθεσία πρέπει να είναι και αναλογική με τον σκοπό και δεν πρέπει να περιορίζουμε τα δικαιώματα περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο. Και κάθε περιορισμός πρέπει να έχει απτή προστιθέμενη αξία. Θεωρείται λοιπόν πως ε, όλα αυτά ισχύουν και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων. Ή μήπως απλά κάνουμε κάτι για να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στίβενς. Ευχαριστώ συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί. Θα περιοριστώ σε μια ερώτηση, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για το έργο των προηγούμενων μηνών. Βλέπω πως στηρίσατε τις προσχέσεις σας και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό τώρα. Η το πρωί διάσα μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χαλβεζέλστραπ που είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας ε, του ΦΕΦΕΝΤΕ στην Ολλανδική Βουλή και είπε πως ε, υπάρχει από ό,τι φαίνεται στην ε, σύμβαση για τους πρόσφυγες η οποία λέει πως έχει κανείς το δικαίωμα σε ασφάλεια στην δική του περιφέρεια του κόσμου αλλά μετά το δεκαετία του 1970 προσθέθηκε το ότι έχει δικαίωμα ασύλου ε, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Ένα πρωτόκολλο προσθέθηκε το 1967 στην ε, σύμβαση του 1951 θεωρείτε πως θα έπρεπε να το εξετάσουμε τουλάχιστον αυτό μου που είτε κάποιο ενδιαφέρον ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ Björk Thank you very much. Um, uh, ευχαριστώ πάρα πολύ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη νομίζω πως ε, δεν υπάρχει λόγος ε, να χαιρόμαστε και ιδιαίτερα Όχι δεν είναι ότι δικιά σας Προεδρία, γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φαίνεται πως ε, δεν έχουμε αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που θα ήθελαν οι πολίτες. Δεν θέλω να επαναλάβω τώρα τις ανησυχίες, τις γνωστές για το ότι μειώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αλλά γεγονός είναι πως όταν μιλάμε για την κατάσταση των προσφύγων που αναζητούν προστασία στην Ευρώπη, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και αυτά που μας λέει η Διεθνής Αμνηστία, η πατερμοσία του ΕΕ τα κτλ. δείχνουν πως γίνεται πιο δύσκολο το φρούριο. Εμεί πήγαμε στα Βαλκάνια, είδαμε την δίωδο τότε από την Ελλάδα, από Γουδουμού και τα Σερβία, στην Κροατία και δεν υπήρχαν διακινητές πριν από 1,5 μήνα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ε, ασφαλή δίδο. Τώρα όμως ακούμε αποθήσεις ότι επανέρχονται ήδη ε, κινητές, γίνεται φιλτεράρισμα στην ε, Πούγουδουμού με βάση την εθνικότητα, οπότε de facto επανήλθαν οι διακινητές, ο κόσμος έχει κολλήσει στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούμε, δεν μπορούμε έτσι να βάζουμε φράχτες. Ε. Κάποιοι το θένε, δεν γίνεται αυτό και είναι και κατά του δικαίου. Οπότε ε, αυτό που λέτε για νέα συνόρια φυλακή δεν έχει καμία δουλειά αν δεν, αν δεν δούμε πρώτα το πώς θα τους υποδεχτούμε και θα τους προστατεύσουμε στην Ευρώπη. Αυτά πρέπει να τα συζητάτε ταυτόχρονα. Πού είναι λοιπόν η συζήτηση για το θέμα της επαναγκατάστασης και τι γίνεται για να καταγγείλουμε αυτά που ακούμε για αποθήσεις στα σύνολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Τζίρεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα οποία είπατε για τους φακέλους που κληρονόμησε η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Γιατί μόνο τότε καταφέραμε να σταματήσουμε το φαινόμενο όταν πολεμήσαμε τους διακινητές. Τώρα για τη Βρετανική ε, πρωτοβουλία. Ήταν ένα ψήφισμα του ΟΗΕ το οποίο αφορούσε μόνο τα ύδατα μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας. Λίγα πράγματα έγιναν λοιπόν. Ειδικά, αν δει κανείς τη Λιβύη, ελάχιστα έχουν γίνει για να σταματήσει ε, η ροή. Δεν θα επανέλθω. Ε, δεν επανέρχομαι για να παραπονεθώ. Γιατί Εντάξει, στο Λουξεμβούργο συντονιστικό ρόλο είχε. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε να δούμε να μας πείτε ποια ήταν τα εμπόδια στην εφαρμογή αυτής της απόφασης. Δεύτερον, μια παρατήρηση. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Μπόνη. Ήταν στην κυβέρνηση, εγώ ήμουν στην αντιπολίτευση και τώρα είναι επικριτικός απέναντι κυβέρνηση την οποία εγώ στηρίζω και πράγματι καλό ήταν το ότι αντέδρασε σε λάθος παρουσίαση των γεγονότων για το τι συμβαίνει στην Πολωνία. Δεν υπάρχουν συλλήψεις. Καλό είναι λοιπόν να προσέχουμε τις επιθέσεις αυτές, ειδικά αφού ο κύριος Σούλτς ε, συνάντησε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σίτβα και ελπίζουμε ότι ενημερώθηκε τελικά ο κύριος Σούλτς για το πόσο λάθος είναι ενημερωμένος. Ε, τέός ομιλητής, η κυρία Λόρενστεν. Ευχαριστώ, Κλοντ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, διότι επειδή ασχολήθηκα με την οδηγία για την προστασία δεδομένων, ε, είχαμε μια πολύ θετική εμπειρία. Αντί να υπάρχει μια μόνιμη διαμάχη μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, ε, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει επικοδομητική συνεργασία. Ένα σαφές ε, χρονοδιάγραμμα από την αρχή ε, είναι αυτό που έκανε η Λουξεμβουριακή Προεδρία. Είπανε ότι είμαστε με τη μεριά του Κοινοβουλίου, έχουμε μία προσέγγιση ε, σε πακέτο, αλλά ο στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα ε, μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Αυτή ήταν μία πολύ καλή αρχή, γιατί υπήρχε ένα σαφές πλαίσιο και σαφές χρονοδιάγραμμα. Και έχω μία ερώτηση τώρα όσον αφορά την εφαρμογή, διότι μετά από αυτή την τόσο καλή εμπειρία, ε, φοβάμαι λίγο για το μέλλον, διότι έχουμε θέσει ένα πάρα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή. Δύο χρόνια για την οδηγία και για τον κανονισμό. Πώς ε, ε, νιώθετε εσείς και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε μια συνεκτική διαδικασία ώστε σε δύο χρόνια να ξεκινήσει όντως η εφαρμογή. Γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Ε, τμήμα αυτού είναι και οι κοινέ ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Κάποιο το ρώτησε. Με αυτές τις κοινέ βάσεις δεδομένων, οι κανόνες που έχουμε καθορίσει αυτή τη στιγμή, τρόπον την να καθορίζουν το πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν πριν έχουμε σαφείς κανόνες για μια πρακτική ανταλλαγή πληροφοριών. Και εδώ έρχομαι στο θέμα των κοινών ορισμών. Είδαμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχουν κοινοί ορισμοί όταν προσεγγίζουμε το θέμα της ασφάλειας. Ε, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν από την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε μια τελική απόφαση για το πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα θέματα ασφαλείας στην οδηγία και έγινε με κάποιους περιορισμούς. Αλλά είναι σαφές ότι προκειμένου να προχωρήσουμε με βάση όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος θα μας λέει πού ε, είναι πραγματικά αρμοδιότητα το κράτους μέλους εθνική ασφάλεια και πού το ξεπερνάει. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ε, για τις κοινέ βάσεις δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών είναι αυτό. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να θίξω. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα θεσμικά όργανα που δεν είναι αποτελεσματικά, την ανάγκη για μια κοινή ε, ε ακτοφυλακή και το καθεξής. Αυτό που λείπει είναι μια πρόταση από το Συμβούλιο. Διότι αυτό είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Η Κομισιόν μας προτείνει κάτι. Το συζητούμε εδώ και μετά το Συμβούλιο ε, μπαίνει σε μια αμυντική στάση και προσπαθεί να μετριάσει τις προτάσεις. Πού είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις του Συμβουλίου, πώς μπορούν πραγματικά να οργαστούν ε, όλοι αυτοί οι θεσμοί που αφορούν τη μετεγκατάσταση, την ε, ε, ακτοφυλακή, γιατί είναι τόσο παθητικό το Συμβούλιο και δεν αντιδρά. Συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που έφυγε ο Υπουργός ε, Μετανάστευσης ε, στα μισά τη συζήτηση, γιατί και κάποιε από τι ερωτήσει στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων σαφώς ε, σχετίζονται με τη μετανάστευση. Νομίζω όμως ότι ο Ετιέν και ο Φέληξ έχουν μια πολύ σαφή εικόνα του τι ακριβώς έκανε η Προεδρία και για τα θέματα της μετανάστευσης. Θα προσπαθήσω λοιπόν, αν θέλετε να σας ζητήσω, αν θέλετε να αφήξετε και τα θέματα αυτά, μπορείτε να αφήξετε και αυτά. Δεν μπορείτε να απαντήσετε βέβαια κάθε ερώτηση, αλλά ως ε, έτσι, οδηγία μπορούμε να το ε, ακολουθήσουμε για να μας απαντήσετε. Μας, έχει περάσει ο χρόνος, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τι έκανε η Προεδρία. Ο Έτια πρώτα. Ευχαριστώ Κλοντ. Θα είναι δύσκολο να απαντήσω σε 7 λεπτά σε ερωτήσεις μιας ώρας, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε δύο ερωτήσεις που ακούστηκαν επανειλημμένως. Ανταλλαγή πληροφοριών ή έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Κάποιοι από εσά το είπαν σαφώς. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπόλ ε, πόρο απέχει από την τελειότητα, επομένως θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο στοιχείων. Αφενός υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και αφετέρου ανταλλαγή αστυνομικών και δικαστικών πληροφοριών. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Λουξεμβουριανή Προεδρία ανέλαβε πρωτοβουλία να προσκαλέσει πέντε υπηρεσίες ε, πληροφοριών στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στα πλαίσια της ομάδας ΚΑΤΣ. Εκεί παρουσιάστηκε η ε, θέση των κρατών μελών και είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια παρουσίαση από το 2001. Ε, ξέρετε ότι αυτό περιορίζεται από τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορεί να είναι διαφορετικοί από τη μία. Και επίσης ε, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Και όπως μας είπατε και εσείς και σας είπα και εγώ στην αρχική μου πρόταση, ε, δεσμευτήκαμε πριν από τον Ιούλιο του 2006 να υπάρχει μια πλατφόρμα Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ε, συνιστά συγκεκριμένο βήμα προόδου. Σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο και εδώ έχουν υπάρξει βήματα προόδου μετά από τις εκκλήσεις που απίθυνε το Συμβούλιο. Πρέπει βέβαια να διαπιστώσουμε ότι πολλά μένει ακόμη να γίνουν έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή ανταλλαγή πληροφοριών που να είναι αντίστοιχη με τη σημερινή απειλή. Είναι λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι μόνο πέντε κράτης μέλη και μία συνδεδεμένη χώρα αυτή τη στιγμή δίδουν το 50% των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο σημείο focal point της Europol. Και μόνο 2.081 μαχητές έχουν καταγραφεί. Αυτό το σημείο επαφής νομίζω ότι είναι ένα βασικό μέσο για την ανείχνευση των κινήσεων των ξένων μαχητών. Οι μισές από τις ε, χώρες δεν ενεργοποιούν το Europol Information System για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουν καταγραφεί εκεί μόνο 1.600 ξένοι μαχητές και οι μισές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει συνδεθεί ακόμα ανάμεσα στις μονάδες που καταπολεμούν την τρομοκρατία ε, και την ε, ε, διασφαλισμένη μορφή επικοινωνίας CNR της Europol. Απαιτούνται λοιπόν νέα μέσα, αλλά ταυτόχρονα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε ήδη στην διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν και κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μια προσπάθεια η οποία έχει σαν σχέση την καταγραφή της κατάστασης ε, έχει ξεκινήσει, κάτι το οποίο θα μας δώσει μια συγκεκριμένη ιδέα για τον μετασχηματισμό και την επεξεργασία των μέσων της Europol, της Interpol και του Eurojust. Σε μια δεύτερη φάση αυτή η καταγραφή της κατάστασης θα εξεταστεί σε βάθος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι νομικά εμπόδια έχουμε και τι τεχνικά εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται παράλληλα να στηρίξει οικονομικά και τεχνικά τα διάφορα κρατημέλη για να καλυφθούν τα κενά τα οποία έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν, όπως η σύνδεση όλων των συνοριακών σταθμών με τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών μέσων έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα τεχνικά εμπόδια για τις διασυνδέσεις. Το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα συστήματα Europol και Interpol. Το κέντρο καταπολέμησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο της Interpol για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας νομίζω ότι θα βοηθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα στηρίξει τις κατασταλτικές υπηρεσίες των κρατών μελών στην επίτευξη των δράσεων τους. Τώρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης είμαστε πεπισμένοι ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε κατασταλτικά μέτρα αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη. Έχουν ξεκινήσει αρκετές πρωτοβουλίες στα πλαίσια μιας στενής συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και τους κοινωνικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Πρέπει να υποστηριχθούν ακόμα περισσότερο με τα διαθέσιμα μέσα της Ένωσης, τα οποία έχουν εξελιχθεί με σημαντικό τρόπο κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Το κέντρο ας πούμε της ε, πρακτικής RIM, ε, Radicalization Awareness Center, ή network μάλλον. Αυτό θα επιτρέψει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από αυτούς που ασχολούνται με το θέμα, από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα του φανατισμού και τους υπευθύνους της κοινωνίας των πολιτών για τα ίδια θέματα. Υπάρχει επίσης και η Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με τα θέματα της Συρίας. Σε, ε, στην εργασίες ε, ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε την δομή αυτή ε, και πέραν του 2016. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πλατφόρμα συνάντησης των κρατών μελών ε, με τις επιχειρήσεις του ίντερνετ όπως η Microsoft, το Facebook, το Twitter. Στόχος αυτού του φόρουμ είναι να βρεθούν κοινέ λύσεις έτσι ώστε να ασχοληθούμε με το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης online. Μετά τις συζητήσεις που έγιναν σε υπουργικό επίπεδο, μία από τις επιχειρήσεις ήδη προχώρησε σε μία τροπολόγηση των συνθήκων χρήσης των μέσων της, για να διευκολυνθεί η απόσυρση του εξτρεμιστικού περιεχομένου στις πλατφόρμες της και να μειωθεί η προπαγάνδα. Το φόρουμ αυτού είναι σε συνεργασία με τη μονάδα Internet Referral Unit που ακολουθεί τις εξτρεμιστικές ε, δράσεις στο εσωτερικό του διαδικτύου και ελέγχεται από τη Europol. Αυτά λοιπόν για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και για τη συγκεκριμένη ερώτηση για τα όπλα, για την οδηγία για τα όπλα, να πούμε ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι πολύ νωρίς. Τώρα παρουσιάστηκε η πρόταση, θα γίνουν ακόμα συζητήσεις και δεν είμαι σε θέση να σας δώσω ήδη από τώρα λεπτομέρειες γύρω από την κατάσχεση των ημιαυτόματων όπλων αλλά είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι το λέτε με κάποια ανακούφιση ότι θα το αναλάβει η Ολλανδική Προεδρία το θέμα. Είναι πολύ περιπλοκόντο το θέμα των πυροβολών όπλων. Φέληξ, ευχαριστώ Κλόμπντ. Καταρχάς να ευχαριστήσω εκείνους που ευχαρίστησαν την ε, Λουξεμβουριανή Προεδρία και θέλησαν να επισημάνουν και το γεγονός ότι είναι οι συνεργάτες ε, οι οποίοι ε, προχωρούν τις εργασίες μέχρι τελευταία στιγμή και θα ήθελα να επισημάνω και αυτό που είπε η κυρία Γκρίσμπεργκ. Ε, όσον αφορά τις διάφορες ερωτήσεις, η κυρία Χολμάιερ επεσήμανε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη στρατολόγηση. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχα και εγώ την ε, ευκαιρία να υπογράψω νομίζω τον Οκτώβριο ξενόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το πρόσθετο πρωτόκολλο το οποίο μεταφέρει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ε, του Σεπτεμβρίου του 2014 για τους ξένους μαχητές και περιλαμβάνει και το θέμα της στρατολόγησης και το γεγονός ότι ε, μπορεί κάποιος να στρατολογηθεί για, για τρομοκρατικές ε, ενέργειες. Υπάρχει λοιπόν μια βάση και η ίδια η Προεδρία πρότεινε ένα κείμενο, μια πρόταση οδηγίας για να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε και στα κρατημέλη το ψήφισμα των ΟΕΕ. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, πρέπει να εφαρμόσουμε τον δίκαιο ενισχύ. Όσον αφορά την πρόληψη, είχα το προνόμιο να διοργανώσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια διάσκεψη στις 19 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες για τις αρχές της πρόληψης ε, στον αγώνα αυτών. Διότι δεν είναι πάντα η καταστολή η οποία προέχει, υπάρχει και η πρόληψη η οποία είναι εξίσου σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι κατασταλτικές ε, δυνατότητες που έχουμε να συνοδεύονται και από αυτό. Και να σας πω ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε ήταν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη συνέχεια και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Τζάι και συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών που ε, καταδεικνύει ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνη και αυτοί ενδιαφέρονται και με τις προληπτικές πτυχές παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά υπάρχει η διάθεση και τα όσα γίνονται είναι πολύ σοβαρά. Ε, δεν είναι εδώ η κυρία που έφτιαξε την ερώτηση και είπε ότι χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη και όχι περισσότερη. Να σας πω ότι εγώ διαφωνώ με την άποψή της. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Η ερώτηση του κυρίου Μπόνι για την ε, συζήτηση ε, αυτή, ναι και αυτό περιλαμβάνεται στα θέματα των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων, διότι είναι τμήμα των νο, μη νομοθετικών προτάσεων και υπήρξε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση στα πλαίσια του Συμβουλίου διότι οι ρητορίες μίσους ε, δεν είναι αποδεκτές, ε, δεν είναι αποδεκτές ούτε στο διαδίκτυο αλλά ούτε στον πραγματικό κόσμο. Και φυσικά υπάρχει νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Ακόμα και αν υπάρχει, υπάρχει διαδικτυακών υπηρεσιών δεν συμμετέχουν στη διαδικασία, ε, όλα τα κράτη-μέλη διαθέτουν νομοθεσία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί. Ε, Σίγουρα δεν μπορεί να διώκονται όλες οι υποθέσεις ε, και να παρακολουθούνται όλες οι υποθέσεις, αλλά στον τομέα αυτό υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και οι εθνικές αρχές δεν χρειάζονται εξουσιοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών για να δράσουν, ε, διότι υπάρχουν δυνατότητες βάση δικαίου. Το Λουξεμβούργο το κάνει τακτικά εδώ και κάποιους μήνες και νομίζω ότι υπάρχουν αντίστοιχες δυνατότητες σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την ερώτηση της Άννας Γκόμες ε, για οικονομικές κυρώσεις που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε. Δεν είναι αυτή η θέση του Συμβουλίου. Δεν εγκρίθηκε κάτι τέτοιο και η Λουξεμβουριανή Προεδρία σίγουρα θα προτιμούσε να υπάρχουν και κάποιες ε, οικονομικές κυρώσεις και να υπάρχει και ένα σύστημα ε, πρημοδότησης αυτών που κάνουν κάποιες προσπάθειες. Ε, τα πρόστιμα δεν θα λύσουν το πρόβλημα, ε, μπορεί να δημιουργήσουν ένα νέο πρόβλημα. Για μένα λοιπόν δεν είναι πανάκια για όλες τις λύσεις και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό είναι πιο επικοδομητικό στη συνέχεια. Θέσατε επίσης και το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Συμφωνώ με την άποψή σας. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει λύση για την νόμιμη μετανάστευση είναι τμήμα του προβλήματος που δημιουργεί πάρα πολλές πιέσεις ε, ε, στις στην παράνομη μετανάστευση. Σίγουρα δεν έχουμε ολοκληρώσει στο θέμα αυτό και δεν έχουμε κάποιες βιώσιμες και εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις, αλλά προσπαθήσαμε στη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας να βρούμε μια λύση, καταλήξαμε σε μια συμφωνία και προσπαθούμε να βρούμε και κάποιες νόμιμες οδούς ε, για να μπορεί κάποιος να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τα πάντα, αλλά έχουμε καταλήξει μια συμφωνία για μια πτυχή που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο κύριος Ντεπρέ ερώτησε κάτι για το τι διαβάζουμε στις εφημερίδες για τη Δανία. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για επίσημη πρόταση της Δανίας αυτή τη στιγμή. Διάβασα και εγώ αυτά που διαβάσετε κι εσείς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για πάγια θέση της Δανίας. Θα περιμένω λοιπόν ε, να το διαβάσω πριν από το σχολιάσω, αλλά συμφωνώ ε, εγώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Αν πραγματικά υπάρξει ε, τέτοια επίσημη πρόταση από τη Δανία θα... Ε, ε, που ασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, συμφωνώ με την άποψή σας. Ε, είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και στο Συμβούλιο Τζάι. Θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής. Πρόκειται για μια πραγματική οδό και συμφωνώ με το αίτημά σας. Η κυρία Κινίτσι αναφέρθηκε στο οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μία από τις πιο επονίδιστες μορφές εγκλήματος, διότι ε, αψηφά το κράτος, αψηφά τις δυνατότητές μας, αψηφά, αψηφά την ηθική μας και δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη μόνα τους να αντιμετωπίσουν μορφές εγκλήματος που ξεπερνούν τα σύνορα και είναι πάρα πολύ οργανωμένες. Και σίγουρα θα πρέπει να γίνει μεγάλη πρόοδος επί του ζητήματος. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα ε, υπήρξε συμφωνία στην οδηγία για την προστασία δεδομένων που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που επιτρέπει και την αντιλαγή πληροφοριών. Και αυτό ε, αφορά κυρίως τις αστυνομικές και δικαστικές πληροφορίες. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών το εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα. Η οδηγία που διαπραγματεύτηκε η συγγήτριά σας, η κυρία Λόρεστιν, ε, μαζί μας θα αποτελέσει θεμέλιο της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών και θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πολύ σοβαρά επί του ζητήματος. Και νομίζω ότι και γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε, διότι συμφωνώ και εγώ με την άποψή σας για το οργανωμένο έγκλημα. Η κυρία Γκρίσμπεργκ έθεσε μια ερώτηση για, την, ε, ε, με τη, για τη διαδικαστική βοήθεια. Ε, Έχουμε ολοκληρώσει δύο θέματα και ακόμα ε, εκρεμεί το τελευταίο. Ε, έχω υπενθυμίσει στους ε, συναδέλφους στο Συμβούλιο ότι δεν είναι θέμα χρημάτων το θέμα αυτό. Σίγουρα θα υπάρχει ένα κόστος για την εφαρμογή του, αλλά ταυτόχρονα θα αξίζει πολλά περισσότερα. Εάν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως κάνουμε τώρα και να εδώ και χρόνια ε, μέσω ολοένα και μεγαλύτερης αμοιβαίας αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις είναι τμήμα τους. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι επίσης αναπόσπαστο τμήμα. Θα πρέπει να τη διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε ε, να έχουμε την πολυτέλεια να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δίνονται τα μέσα ώστε να μπορούν κάποιοι να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν είναι λοιπόν μόνο ένα κόστο, είναι μια διαδικαστική εγγύηση που είναι ικανή και αναγκαία στη συνθήκη για την ε, αμοιβαία αποδοχή δικαστικών αποφάσεων. Το υπενθύμησα επανειλημμένο στο συναδέλφους και ελπίζω ότι η Ολλανδική Προεδρία θα συνεχίσει τη συζήτηση για αυτό το τρίτο κείμενο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να ε, επιτρέπεται σε όλους τους πολίτες μας να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα με το που διαμένουν, είτε στη χώρα καταγωγής τους, είτε σε κάποια άλλη χώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το κείμενο και ως Υπουργό Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου που ε, σύντομα θα έχει και ελευθερία λόγου ε, θα συνεχίσω να πιέζω για αυτό το ζήτημα. Η κυρία Κάουφμαν αμφισβήτησε την αισιοδοξία μου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, το είπα για να ενθαρρύνω και τους συναδέλφους από την Ολλανδία που χρειάζονται και αυτή μεγάλη ενθάρρυνση και υπομονή και επιμονή σε αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνικό ε, εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκαν τα άρθρα από το 1 έως και το 35 και πολύ σύντομα, αύριο νομίζω ή μεθαύριο η Λουξεμβουργιανή Προεδρία θα δημοσιεύσει ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει το ε, κείμενο των άρθρων 1 έως 35, το οριστικό τα οποία έγιναν ε, στη διάρκεια της τριάδας των Προεδριών, στο Τρίο και όχι μόνο στη Λουξεμβουργιανή Προεδρία, θα δημοσιευθεί αύριο και θα είναι δημόσιο λοιπόν έγγραφο. Μπορείτε να δείτε τα άρθρα 1 έως και 35, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε και τη συζήτηση με την Ολλανδική Προεδρία η οποία θα είναι εδώ, όπως είπε και ο πρόεδρος ράζ, από τις 11 Ιανουαρίου. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουμε αυτό το κείμενο. Η κυρία Στίβεν έθεσε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για δύο μέσα του διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς δεν τα γνωρίζω επαρκούς, επαρκώς. Ε, πρόκειται για αρμοδιότητα του συναδέλφου Άσεμπορκ που χρειάστηκε να φύγει. Επομένως δεν μπορώ να απαντήσω ε, στην ερώτησή σας, ζητώ συγγνώμη τελευταία ερώτηση ήταν, ε, ήταν η κυρία ε, Λάουρεστεν, ο οποίος έθεσε αρκετές ερωτήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία δεδομένων και του σχετικού κανονισμού. Ξέρω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ε, προετοιμάζουν την ενεργοποίηση της οδηγίας. Έχουμε δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα και η Προεδρία φυσικά ε, πρέπει να πιέσει τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη μεταφορά του κειμένου και την, ε, στην εθνική του νομοθεσία, αλλά υπάρχουν κίνητρα και για τα κράτη-μέλη. Τελευταία ερώτηση αφορά τη μετεγκατάσταση, το relocation. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σε επίπεδο Συμβουλίου ενεργοποιήσαμε τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του μηχανισμού EPCR για τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό αποφασίστηκε επισήμως στο Συμβούλιο προς τα τέλη του έτους και μετά από αυτό έγιναν αρκετές συνεδριάσεις ε, παρακολούθησης παρουσία των Ιταλών, ε, Ελλήνων και Τούρκων συναδέλφων ε, και άλλων. Και από όλα αυτά έχει ε, ε, εκπονηθεί μια έκθεση που συζητήθηκε στο Συμβούλιο και είναι δημόσια. Επομένως δραστηριοποιηθήκαμε και σε αυτό. Αυτή ήταν η τελευταία μου παρατήρηση και θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας όλους για την εξαιρετική συνεργασία αυτό το εξάμεινο και ε, χαίρομαι που θα σας ξαναδώ από εδώ και πέρα με την ιδιότητά μου ως Υπουργός του Λουξεμβούργου και όχι ως Προεδρεύων του Συμβουλίου. <clears throat> Thank you, Felix. Um, Σας ευχαριστώ Φίλιξ, ευχαριστώ Ετιέν. Όπως γνωρίζετε είναι η τελευταία επίσημη επαφή μας ε, με τους υπουργούς του Λουξεμβούργου. Μας περιμένουν στις 11 Ιανουαρίου οι Ολλανδοί υπουργοί. Αλλά νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα και η σωστή στάση των Λουξεμβουργιανών υπουργών που ήσαν τουλάχιστον εδώ σήμερα αντιμετώπισαν τις προκλήσεις υπαρξιακού τύπου κάποιες από αυτές και σε μια πρώτη επαφή γνωριμίας οι Ολλανδοί Υπουργοί είπαν ότι το παράδειγμα που έδωσαν οι Λουξεμβούργοι είναι ένα σωστό αλλά και δύσκολο παράδειγμα. Τίθεται το θέμα το πώς τα ευρωπαϊκά όργανα θα αντιμετωπίσουν τα θέματα είναι ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε ε, τις χρονικές προθεσμίες ε, για κάποιες διαδικασίες νομοθετικές που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι Λουξεμβουργιανοί υπουργοί στη συμμετοχή τους στον τριγωνικό διάλογο πέτυχαν πάρα πολλά. Ήταν μια προεδρία που συγκέντρωσε την προσοχή της και στα θέματα της δικαιοσύνης. Ήταν εκεί και ο κύριος Μπόνι ήταν μια διάσκεψη ουσιαστικά που εμείς συνδιοργανώσαμε και μπορέσαμε μαζί με σας και με τα υπόλοιπα μέλη εδώ να συνεργαστούμε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα με σωστό τρόπο. Έχουμε πολλούς ε, στόχους να πετύχουμε τους επόμενους έξι μήνες, ε, πολλές εφαρμογές ηλιμένων αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πάντως για την προσπάθειά σας μέχρι τώρα και προσβλέπουμε στη σωστή συνεργασία και με τους διαδόχους σας. Ευχαριστώ πολύ. Colleagues, um, uh, Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει συνάδελφοι. δώσαμε σε όλους το λόγο γιατί ήταν πολλοί συνάδελφοι και οι εισηγητές που συμμετέχουν επίσης και στους τριμερείς διαλόγους. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση λοιπόν. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, δημιουργία του Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, την κυρία Ιντβελτ πρώτα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη γιατί οι περισσότεροι παρόντες θα γνωρίζουν τα της έκθεσης. Πρόκειται για έκθεση νομοθετική πρωτοβουλίας που ζήτησε η Ολομέλεια για να αναπτυχθεί ένα μηχανισμό για να διαφυλάξουμε το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και νομίζω πω η ανταλλαγή απόψεων κατέδειξε την ανάγκη ενός τέτοιου μηχανισμού γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίε αρχέ στη συνθήκη στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, νομολογία κτλ. Αλλά βλέπουμε όλοι πως ε, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία περνάνε καιρούς δύσκολους. Οπότε χρειάζεται ένας μηχανισμός ε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε μια κοινότητα αξιών όπως θέλουμε να είμαστε. Έχουμε συναντηθεί ήδη δύο φορές με τους σκιώδεις εισηγητές ε, για μια γνωμοδότηση και για τη ΣΑΦΚΟ γιατί θέλουν να συνεργαστούμε ως μια ομάδα πέρα από τα, τους επίσημους κανόνες. Και βεβαίως τα διαχωρίσαμε αυτά. Δηλαδή κάναμε ένα καταμερισμό εργασίας μεταξύ μας. Κάθε λοιπόν σκιώδης συγητής ε, και ο συγητής της ΑΦΚΟ θα προετοιμάσει ένα έγγραφο εργασίας το οποίο θα σας προτείνουμε στα μέσα Φεβρουαρίου. και μετά ελπίζουμε να πάμε μέχρι τον Ιούλιο στην Ολομέλεια βεβαίω αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο νομίζω πως πρέπει να καθυστερήσουμε λίγο για να έχουμε κάτι το θετικό το οποίο θα αγκαλιάσουν όλοι αντί να είναι κάτι το επίμαχο τα έξι θέματα θα είναι πρώτον ο πίνακα βαθμολογία για δημοκρατία, κράτο δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Δεύτερον, η, δεύτερη πανε, η ετήσια πανευρωπαϊκή κοινοβουλευτική συζήτηση. Τρίτον, μια αξιολόγηση αντικτύπου η διαδικασία ελέγχου. Τέταρτον, η χρήση του άρθρου 2 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως ε, βάση για διαδικασία παραβάση. Πέντε, ατομική, ε, αν μπορεί να είναι ένας μηχανισμός τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν μεμονωμένοι πολίτες και έκτον υφιστάμενοι μηχανισμοί. Για το τελευταίο θέμα, υφιστάμενοι μηχανισμοί, θα κάνουμε, είχαμε μάλλον μία μικρό ακρόαση πριν από 15 μέρες και σκοπεύουμε να κάνουμε άλλη μία στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με την ΑΦΚΟ με τους εκπροσώπους ε, της δικαστικής εξουσίας ε, του ΔΕΚ, ίσως συνταγματικών δικαστηρίων από τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε και από τη ΣΥΠΑ γιατί έχουν περισσότερη εμπειρία με αυτά τα ζητήματα. Οπότε θα είναι ενδιαφέρον. Και βέβαια θα συναντηθούμε και με το Συμβούλιο και την Προεδρία. Ακούσαμε σήμερα και από του Λουξεμβούργιου ότι είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και ήταν μια αρχή συγκρατημένη και ελπίζουμε η Ολλανδική Προεδρία και οι επόμενες να την αναπτύξουν. Και ελπίζω αυτό να γίνει από κοινού Συμβούλιο, δηλαδή Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Αυτά. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίε, μπορώ να σας στείλω email. Ευχαριστώ. Πρόκειται λοιπόν για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το έγγραφο εργασία θα παρουσιαστεί 15 και 16 Φεβρουαρίου στη Λίμπε και θα γίνει και μία μήνυα ακρόαση με την ΑΦΚΟ στι 22 Φεβρουαρίου. Έχοντα λοιπόν αυτά κατά νου, α ακούσουμε τους και οδησίγητες ε, Ευχαριστώ. Κλοντ. Αυτή τη φορά δεν θα μιλήσω ε, Λουξεμβριανό. Θα ήθελα να πω το εξή. Το ίδιο με πριν, δηλαδή. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, από τη σκοπιά του ΕΛΚ είναι κέριο για την έκθεση αυτή και πρέπει να προσέξουμε το θέμα πρέπει να αφορά όλες τις ίδιες λεπτομέρειες ε, που μας απασχόλησαν και την άλλη φορά για μια χώρα στον κέντρο της Ευρώπης ε, γιατί παρόμοια πράγματα μπορούμε να βρούμε ουσιαστικά για κάθε κράτος μέλος αλλά πρέπει να προσέξουμε να δούμε αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή λογική διακυβέρνησης ε, που είτε έχει ήδη επιτευχθεί είτε θεωρούμε πως πρέπει να επιτύχουμε. Και αυτό σχετίζεται με το κράτος δικαίου, με την προβλεψιμότητα του κράτους, με την αξιοπιστία του κράτους και με όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Και βεβαίως με τη διάκριση των εξουσιών, ανεξάρτητη δικαιοσύνη κτλ. Και πολλά από αυτά τα πράγματα είτε υφίστανται επιθέσεις είτε δεν λειτουργήσαν ποτέ, αν δούμε το τι σημαίνει τώρα στην Ελλάδα. Όχι μόνο η χώρα αυτή δεν ελέγχει ακριβώς τα σύνορά της, κατόπιν είναι πρόβλημα και για την ίδια και για την ζώνη Σέγγεν, αλλά υπάρχουν και εσωτερικά ζητήματα, Εφόσον αυτή η χώρα σε πολλά μέτωπα ποτέ δεν είχε επιτύχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είτε μιλάμε για απουσία διαφθοράς, για αξιοπιστία της διοίκησης, για λειτουργία της διοίκησης και ό,τι σημαίνουν όλα αυτά. Παλαιά φαινόμενα, καινούργια φαινόμενα, αλλά φαινόμενα που βρίσκονται παντού. Και βεβαίω αυτά τα οποία έχουμε τώρα με την τρομοκρατία που μπορούν να μας πάνε, να μας εκτροχιάσουν αν δεν προσέχουμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και πρέπει να είμαστε άρα κάπως ε, προσεκτικοί για να συνεισφέρουμε κάτι ουσιαστικό. Ε, πρόεδρε. μία και καλή στο τέλος, λέει ο πρόεδρος. Έκανα, έκανα λάθος, ε, λέει η κυρία Νετφέλτ, το ξέχασα αυτό. Είναι και αυτό θέμα ενός εγγράφου εργασίας και ζητώ συγγνώμη. Δεν δεν ήθελα να το πω, δεν ήθελα να το πω. Ε, ναι, ναι, κοιτάξτε, ζήτησα συγγνώμη, Χριστούγεννα είναι. Μια φορά το χρόνο το κάνω. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, κύριος Χιακόπ. Κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Νομίζω ότι μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι ότι καταλήγουμε μόνιμα σε μια κατάσταση όπου η εφαρμογή αρχίζει να εξετάζεται μόνο εφόσον καθίσταται προβληματική και δεν την εξετάζουμε την αρχή της περίοδου εφαρμογής ενός μέτρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δικαστής, εμείς δεν είμαστε. Θα θέλαμε να δούμε τα κράτη-μέλη να συμφωνούν με τις βασικές αρχές και να παρακολουθούνται σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των, βασικών αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσφατα υπήρξαν και εκφράστηκαν ανησυχίες από ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου σε σχέση με μεμονωμένες χώρες. Μερικές φορές αυτό είναι κάτι το αντικειμενικό, μερικές φορές ε, ειλικρινά είναι αυστηρά πολιτικό και υποκειμενικό. Οι βασικοί κανόνες, αυτοί καθεαυτοί, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθορίζονται, είναι αντικειμενικοί, αλλά αυτή τη φύγουμε από την αντικειμενικότητα, τότε νομίζω ότι χάνουμε από μπροστά μας τα πραγματικά γεγονότα και το τι πραγματικά συμβαίνει τίθεται λοιπόν ένα θέμα, θα πρέπει να είμαστε πολύ διστακτικοί ε, ονοματίζοντας με, με, χώρες ε, και καταστάσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, πάρα πολλές παραβιάσεις κάποιων κριτηρίων σε πολλές χώρες, όλες σχεδόν οι χώρες, κάτι παραβιάζουν. Και όμως αντί να υπενθυμίσουμε ακριβώς την κατάσταση αυτή και να τους πούμε εξ αρχής να φανούν προσεκτικοί, τότε πραγματικά περιμένουμε ένα σκάνδαλο τεράστιο να φανερωθεί από τα μέσα ενημέρωσης και μετά επιτιθέμεθα στη συγκεκριμένη χώρα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν μου φαίνεται λογικό. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να επανακάμψουμε στις βασικές αρχές μας στην κατάλληλη αντίδραση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας, η Επιτροπή έχει τη συγκεκριμένη ευθύνη για την εφαρμογή και μην εγκαταλείπετε το θέμα αυτό, μην αγνοείτε το θέμα αυτό και μην ασχολείστε με αυτό μόνο αφού πολιτικοποιηθεί και αντιμετωπιστεί με πολύ υποκειμενικό τρόπο. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια για την πλήρη συμμετοχή των σκιωδών από την αρχή των εργασιών και να εκφράσω δύο σκέψεις σχετικές και με τη χάρτα και με το άρθρο 2 με το οποίο ασχολήθηκα σαν σκιώδης εισηγήτρια. Καταρχάς η εμβέλεια Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με τις ε, προβλέψεις του άρθρου, ιδιαίτερα στο άρθρο 51, περιορίζουν τις δυνατότητες ε, εφαρμογής. Νομίζω ότι πρόκειται για αναφορές ε, στον τρόπο με τον οποίο έχουν δεσμευτεί οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ιουσδήποτε περιορισμού στην πλήρη εφαρμογή του, χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεύτερον, περνάω στο άρθρο 2. Αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα ενός αποτελεσματικού σχετικά με τα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν όμως στο μέλλον το θέμα αυτό να συμπεριλαμβάνει όλους όσους συμμετέχουν σε διαδικασίες κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θεσμικά όργανα, χώρες και όσους όσους δρούν στην περιοχή αυτή. Τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της χάρτας είναι ουσιαστικά ο σκελετός πάνω στον οποίο βασίζεται η δράση της Ένωσης και επιτρέπει μια ενισχυμένη συνεργασία που επιτρέπει να ξεπεραστούν τα αντίστοιχα άρθρα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την πρώτη φράση, έχει φάσει, συγγνώμη, έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι ο μελλοντικός μηχανισμός προστασίας δεν θα πρέπει να αναπαράγει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή του 7 σε επίπεδο διακυβερνητικό, όπου περιλαμβάνεται με άλλα λόγια ο κεντρικός ρόλος των νομοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα πιο κατάλληλα να ορίσουν το δίκαιο λόγω της φύσης τους και της προνομιούχας σχέσης με το αντικείμενο. Η απουσία ή ασδήποτε αναφορά σε κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι που τίνει να μετασχηματίσει το νέο μέσο σε μια απλή αναπαραγωγή του άρθρου 7. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω έναν έλεγχο. Έχουμε δύο ομιλητέ, ο κύριο ε, Λόπεθ Αγγιλάρ και μετά κυρία Φαζόν και θα κλείσει ο κατάλογο των ομιλητών αν δεν σα πειράζει. Θα είμαι σύντομο γιατί δεν είναι σχόλιο, ερώτηση είναι. Ναι, συγγνώμη. Εσένα, εσένα, ναι, σε εσένα ήθελα να δώσω το λόγο. Λοιπόν, θα είμαι σύντομο γιατί δεν είναι ερώτηση, είναι σχόλιο, ε, μάλλον δεν είναι σχόλιο, είναι ερώτηση. Ένα δείκτη τη ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην ευρωπαϊκή νομική κουλτούρα εδώ και χρόνια ήταν ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο ε, Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και οι καταδίκες κάποιες χώρας από το δικαστήριο. Ε, ορισμένες φορές είχαμε ε, αλματώδη αύξηση κάποιων συγκεκριμένων χωρών ε, τα τελευταία χρόνια και αυτό μας δείχνει πώς έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς έχει επιδεινωθεί και πώς το βίωσε αυτό. Ε, υπήρξε και μια μεγάλη διεύρυνση φυσικά του δικαστηρίου. Ε, φτάσαμε στις 47 χώρες και πολλές από αυτές δεν είχαν δημοκρατικό ε, υπόβαθρο. Υπάρχει δυνατότητα να προβλέψουμε και ένα μηχανισμό ε, ε, για το ρόλο που θα διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων στις περιπτώσεις τις οποίες είναι ουσιαστική ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι υπάρχουν κάποιες υποθέσεις πολύ σημαντικές, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, το δικό μας το δικαστήριο, άρχισε να αξιολογεί και να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ε, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράμετρο για να αξιολογήσει ε, κατά πόσον τηρούν το κράτος δικαίου τα κράτη-μέλη βάσει του νέου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορούμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ. Η Τάνια Φαϊζόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό και πολύ συχνά στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί στις δυσκολίες σε αρκετά κρατημέλη και στην Ουγγαρία αλλά και σε άλλες χώρες. Και πέραν του πολύ ευαίσθητου άρθρου 7 δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να μας επιτρέπει να δράσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσεις τους ε, τίτλους του εγγράφου εργασίας και νομίζω ότι σε αυτό το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι να έχουμε ένα κατάλογο δικτών. Νομίζω ότι αυτή είναι η, πρόταση, πρόθεση των εγγράφων εργασίας για να ξέρουμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε ε, το επίπεδο της δημοκρατίας στις χώρες μας και επίσης θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και σαφής στόχος να αναπτύξουμε κάποια εργαλεία και μέτρα για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Ίσως ε, θα μπορούσε να μας πεις και δύο λόγια παραπάνω ε, ως προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε όταν υπάρχει παραβίαση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ε, και φυσικά έχει όλη μας την υποστήριξη γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι κρίσιμη σημασία στους επόμενους μήνες και χρόνια. Ε, κύριε Γέρεκ, είχατε φύγει, σας είχα διαγράψει από τον κατάλογο, αλλά να σας δώσω το λόγο ως τελευταίο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη ερώτηση που ακούστηκε. Θα ήθελα κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για το νομικό μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βάσει αυτού του νέου μηχανισμού. Τι διαφορά έχει από τις ε, νομικές διατάξεις ε, των συνθήκων. Και τι διαδικασίες θα ενεργοποιούνται η ερώτησή μου δηλαδή είναι ποια είναι τα καινούργια στοιχεία σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Σόφη, έχουμε καθυστερήσει 20 λεπτά και περιμένουν οι συνάδελφοι για το επόμενο θέμα. Ζητώ συγγνώμη. Ε, πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, επομένως δώσε απλώς μια άγουσα. Ε, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη, θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έχουμε δεν θα είναι ένα νομικό μέσα, θα ε, είναι μάλλον ένα σύνολο μέσων τα οποία θα αποτελούν ε, μαζί ένα μηχανισμό. Και νομίζω ο Τίμωθη πέτυχε ακριβώς το στόχο όταν είπε ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η πρόληψη. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώς στα κρατημέλη. Ο μηχανισμός λοιπόν θα πρέπει να λειτουργεί βαθμιδών μετά από το διάλογο με το, ε, το Συμβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να είμαστε στο πρώτο στάδιο και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια προειδοποίηση για παράδειγμα και μετά θα φτάνουμε στις κυρώσεις είτε είναι το άρθρο 7 είτε είναι κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι να μην ξεχωρίζουμε κάποια χώρα, να μην περιμένουμε να ξεσπάει κάποιο μεγάλο ε, σκάνδαλο αλλά να υπάρξει μια νοοτροπία ε, να εμπεδώσουμε αυτή τη, το θέμα του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις περιπτώσεις που έχει σημασία ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό θα καλύπτεται ε, εκτεταμένα. Θα καλυφθεί τουλάχιστον ελπίζω στι 22 Φεβρουαρίου όταν θα γίνει η ακρόαση με εκπροσώπους του δικαστικού ε, σώματος και μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Τέλος προς την Τάνια Φαγιόν να πω ότι ναι, συμφωνώ ότι η ανάπτυξη δικτών είναι πολύ σημαντική. Το πώς θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον βέβαια θα δούμε. Αλλά είναι και αυτό που είπε και ο Φρανκ Έγγελ. Πώς ορίζουμε τη δημοκρατία, πώς ορίζουμε το κράτος δικαίου και πώς τα μετράμε, με, βάση ποια πρότυπα. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Τίμερμανς μέχρι τώρα αρνήθηκε να ε, προχωρήσει σε προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορεί βέβαια να υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε ε, τη μέτρηση πιο απτή. Το κάνουμε για χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς αξιολογούμε αν πληρούν τις προδιαγραφές, επομένως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προδιαγραφές και να τις ορίσουμε και για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Έτσι, όπως είπε και ο Τίμωθη, θα αποφύγουμε μάλλον και αυτή την πολύ πικρή και ανούσια διαμέχη για την τάδε τη δίνα χώρα ή το τάδε το δίνα πολιτικό κόμμα. Και πρέπει να σου πω, σας πω ότι μέχρι τώρα έχω πολύ απογοητευτεί γιατί έχουμε κάνει ελάχιστα για τη βελτίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ελπίζω ότι στη διαδικασία εκπόνησης αυτής της έκθεσης και στο βασικό αίτημα ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει νομοθετική πρόταση θα αποτελέσει και μια ε, εκκίνηση ώστε να υπάρξει μια πραγματική υλοποίηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 5 στην κατάσταση στη Μεσόγειο και στην ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση προς τη μετανάστευση. Έχουμε δύο έγγραφα εργασίας από τις συντάκτρες, την κυρία Ρομπέρτα Μάτσολα και την κυρία Κιέγγε. Ε, διαχείριση συνόρων και πολιτική θεώρηση των και ο ρόλος της Φρένταξ και των άλλων σχετικών ε, υπηρεσιών, η ε, αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη μετανάστευση και το ρόλο της ε, υπηρεσίας ασύλου. Δεν θα κάνω εισαγωγέ και θα περάσουμε στην παρουσίαση του πρώτου γράφου εργασία για τη διαχείριση των συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων. Μετά από την παρουσίαση του κάθε εγγράφου θα σας δίνω το λόγο για ερωτήσει και να ευχαριστήσω του συναδέλφου που έμειναν και περίμεναν παρά την καθυστέρηση σήμερα το απόγευμα. Η κυρία Μέτσολα θα λάβει πρώτα το λόγο. Ε, απλώς ε, πέστε μου θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση. Τώρα, να δώσουμε πρώτα το λόγο νομίζω στη Ρομπέρτα Μέτσολα. Θα αναφερθεί στο πρώτο έγγραφο εργασία για τη διαχείριση συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ναι, για να μην καθυστερούμε. Θα κάνω μία εισαγωγή για όλα τα έγγραφα και θα είμαι σύντομη πλησιάζουμε το τέλος μιας επίπονης διαδικασίας καθώς παρουσιάζουμε τα τελευταία έγγραφα εργασίας δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα αλλά πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ των διάφορων πολιτικών ομάδων σε ένα θέμα το οποίο πολλώνει ξεκινήσαμε πως ε, για να έχουμε μια ενιαία απάντηση στη μετανάστευση θα χρειαζόταν μια γενική προσέγγιση που θα εξέταζε κάθε πτυχή του θέματος. Βρήκαμε 8 τομείς ε, που έπρεπε να εστιάσουμε και σήμερα παρουσιάζουμε τους τελευταίους, τα σύνορα και την νόμιμη μετανάστευση. Ε, για τα σύνορα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε πως για να μην υπάρχουν εσωτερικά σύνορα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και βέβαια να μοιραζόμαστε πληροφορίες ειδικά μέσω του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Το ένα πρέπει να αντισταθμίζει το άλλο. Η ακαιρεότητα της ζώνης ε, Σέγγεν και η κατάργηση των εσωτερικών σύνορων εξαρτάται από το να, έχει, από να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών σύνορων με υψηλέ προδιαγραφέ που εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα. Η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων θα διασφαλίσει μια οργανωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη και ασφάλεια για όσους χρειάζονται προστασία. Ιδιαίτερα η σωστή καταγραφή και ταυτοποίηση ανθρώπων, ανθρώπων που χρειάζονται προστασία αλλά και η απαραίτητη έλεγχη ασφαλείας. Αναφέρουμε λεπτό, μέρο το τι θέλουμε από την Frontex και βεβαίως τι άποψη έχουμε για την νέα προτινόμενη υπηρεσία που θα ασχοληθεί με την διαχείριση των συνόρων, ειδικά με βάση την κατάσταση που υπάρχει του τελευταίου μήνε, μια αποτελεσματική στρατηγική του τελευταίου μήνε για τη διαχείριση των εξωτερικών μα ε, συνόρων και τη διασφάλισή του, είναι αναγκαία και αναμένω βεβαίω και τι διαβουλεύσεις για την πρόταση τη Κομισιόν. Το δεύτερο έγγραφο εργασία αφορά το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Αυτό ήταν δύσκολο ειδικά όταν μιλάμε για το Δουμπλίνο, πρέπει να αντιληφθούμε τους περιορισμούς του και το γεγονός πως είναι σαφές πως τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα, έτσι ώστε η Ευρώπη να έχει ένα ενιαίο σύστημα ασύλου. Καταθέτουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις για την αναθεώρησή του. Για το θέμα της μετεγκατάστασης όταν ο κόσμος φτάνει στην Ευρώπη και χρειάζεται προστασίες, ακριβώς φτάνει στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να μοιράζονται τις ευθύνες και όχι μόνο αυτά που είναι στα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει αυτό να αποτελέσει πυλώνα οποιασδήποτε αλλαγή ε, στους νόμους ασύλου. Μιλάμε για το Eurodac. Και το γεγονός πως το άρθρο 9 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δακτυλοσκοπούν ε, όλους τους ετούντες άνω των 14 ετών. Επίση υπάρχει ένα έγγραφο για την νόμιμη να γνωρίζουμε πως για να σταματήσει ο κόσμος να έρχεται παράνομα με σάπιο κάραβα και όταν φτάνουν τελικά να τους επιστρέφουμε ε, δεν είναι κάτι το μακροπρόθεσμο αλλά σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα κάθε κράτος μέλους να καθορίζει τον αριθμό των υπήκων τρίτων χωρών είναι και θα πρέπει να συνεχίσει να παραμένει βασική αρχή της οποιασδήποτε προσέγγισης. Μιλάμε λοιπόν για την μπλε κάρτα και ζητάμε η μεταρρύθμισή της να είναι και στοχευμένη και φιλόδοξη και να βρουν τα κατημέλη τα κενά στην αγορά εργασίας όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν επικόδους των χωρών. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι τομείς μπορούν να βελτιωθούν. Και τα επόμενα βήματα τώρα είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έγγραφα εργασίας και άλλες μελέτες και τα ψηφίσματα που έχουμε εγκρίνει μέχρι στιγμής και θα δουλέψουμε τα Χριστούγεννα για να προετοιμάσουμε μια έκθεση που θα σας παρουσιάσουμε στις 18 Ιανουαρίου όπως είπα. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, αντιλαμβάνω πως κάποιοι συνάδελφοι δυσκολεύονται να συνυπογράψουν εκθέσεις με εμένα και την Σεσίλια και εγώ θα ήθελα να σου πω να προτείνουν τροπολογίες. Όμως πρέπει να πω πως θεωρώ πως ε, αυτό το σχέδιο των εγγράφων προκύπτει ε, από την μέγιστη δυνατή διακομματική στήριξη. Και βλέπουμε πως δεν μπορεί βέβαια ο καθένας να παραμείνει στις θέσεις που είχε μέχρι τώρα το κόμμα του. Τώρα πριν στο λόγο Σεσίλια να σας ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη και τη συνεργασία και την ενότητα. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αν είναι να κάνουμε κάτι. Και καλά Χριστούγεννα εύχομαι και καλή χρόνια. Ευχαριστώ. Να έπρεπε το πω στην αρχή. Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις 18 Ιανουαρίου για την έκθεση αυτή ε, γιατί για το θέμα της μετανάστευσης ε, είναι πολύ πολιτικό το ζήτημα, δεν θα είναι εύκολο. Η τελευταία συζήτηση λοιπόν πριν την παρουσίαση της έκθεσης στις 18 Ιανουαρίου. Η Σεσίλ θέλει να προσθέσει κάτι ως συνεισηγητρία. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την ολοκλήρωση αυτών των τριών εγγράφων εργασίας μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε την προπαρασκευαστική δουλειά στο σχέδιο έκθεσης το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί όπως είπε η συνάδελφος και θα φτάσει στην Ολομέλεια στις 18 Ιανουαρίου. Όπως είδατε τα έγγραφα είναι λεπτομερέστατα, δείχνουν την σημερινή κατάσταση περιγράφουν το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, περιλαμβάνουν τις μελέτες και τις απόψεις που ακούστηκαν μέχρι τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις των σκιωδών εισηγητών και εισηγητριών και προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια συμβιβαστική λύση με όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ την Μετσόλα λοιπόν, την συνάδελφο Μετσόλα για τη διαθεσιμότητά της και όλους τους σκιώδεις που έχουν συνεισφέρει στην ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο περιεχόμενο αυτών των τριών εγγράφων, ξεκινώντας από το κοινό σύστημα ασύλου με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κανονισμός αυτός δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει το πνεύμα ε, μέσα από το οποίο δημιουργήθηκε γρήγορη πρόσβαση δηλαδή στη διεθνή προστασία και βελτίωση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, αποφεύγοντας το asylum shopping. Ιδιαίτερα με τις έκτακτες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων χρόνων, οι διαδικασίες του Δουβλίνου είναι περίπλοκες, φαραωνικές θα έλεγα, κοστίζουν, τα κριτήρια που εφαρμόζονται, εφαρμόζονται πολλές φορές αυθαίρετα, παρά την ιεράρχηση από πλευράς του κάθε φορά αρμόδιου κράτους μέλους των διαδικασιών. Προβλέπεται καταρχάς η ύπαρξη οικογενειακών θεσμών, ενώ το κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι το της πρώτης εισόδου. Η παρουσία αποτελεσματικών δεσμών με μία ή περισσότερες χώρες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση και με τον τόπο πρώτης εισόδου, που πολλές φορές καθορίζεται με υποχρεωτικό δεσμευτικό τρόπο από τους σωματέμπορους και από τη γεωγραφία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν μια κοινή ερμηνεία του όρου συγγενικές σχέσεις που να ξεπερνούν τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Η Επιτροπή στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού θα πρέπει να περιγράψει τα όρια τα οποία έχει συναντήσει και να προτείνει φιλόδοξα προγράμματα. Ένα κεντρικό, πολυσυλλεκτικό αν θέλετε κέντρο για, ε, ε, ε, για τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και της ευθύνης από όλα τα κράτη-μέλη. Ανώτατα όρια ανακράτος μέλος, πέρα από το οποίο θα προβλέπονται διαδικασίες ε, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τις αντίστοιχες των υπολείπων κρατών μελών. Αυτό που ζητάμε είναι μια περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών υποδοχής σε όλη την Ευρώπη για να αποφύγουμε τους λεγόμενες δευτερεύουσες κινήσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι θετικές, αλλά πολλά είναι τα κρατημέλη που δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία λέει το σύστημα και δεν τα συμπεριλαμβάνουν στο εθνικό του σύστημα. Αυτό εμποδίζει την εκτίμηση για τα θετικά και τα αρνητικά του συστήματος. Τώρα, για την οικονομική μετανάστευση και τα κανάλια οικονομικής μετανάστευσης, εδώ βασιζόμαστε στην παρούσα συγκυρία το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο ασχολείται με τα θέματα της εισόδου εκπροσώπων ή πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, που δημιουργούν θα έλεγα ε, μια εικόνα σε σχέση με μια Ευρώπη η οποία δημιουργεί, έχει προβλήματα δημογραφικά και στον τομέα της απασχόλησης και το κεφάλαιο των μεταναστών δεν χρησιμοποιείται σωστά και θα υπάρξει μια ανησυχητική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το 2020. Και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί επαναλαμβάνω ότι το 70% αυτών που έρχονται στην Ευρώπη δεν έρχονται σαν οικονομικοί μετανάστες. Το σύστημα είναι ε, ε, σε κατάσταση πολυδιάσπασης και δεν λαμβάνει υπόψη μια συνολική αντιμετώπιση των ε, διαφορών στις αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουν τα όρια των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε στο μέλλον να έχει γενικούς ενιαίους κανόνες η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική μετανάστευση συστήνουμε μια καλύτερη διαδικασία αναγνώρισης των ικανοτήτων των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορούν οι μετανάστες να κάνουν ε, δουλειές αντίστοιχες με τις ικανότητες τους. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέα μέτρα και ενωτόμα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τώρα για την μπλε κάρτα. Εγώ δεν θεωρώ ότι το μέσο αυτό είναι στο ύψος των περιστάσεων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να θεωρηθεί σαν κανάλι νόμιμης μετανάστευσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να διασφαλίσει να μην υπάρχουν αντιθέσεις με τα εθνικά συστήματα. Αυτό το οποίο ελπίζουμε είναι μια αναθεώρηση της οδηγίας φιλόδοξη ιδιαίτερα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής. Τέλος, το τελευταίο ε, έγγραφο εργασίας είναι η πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων. Όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε και εμείς να λάβουμε υπόψη μας το ότι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων είναι τμήμα της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Ζητάμε γι' αυτό λοιπόν την σωστή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται από το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και στα σημεία εισόδου και στα σύνορα γενικότερα και στα πλαίσια του ελέγχου των εθνικών υδάτων ε, και ε, φυσικά στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και διάσωσης. Νομίζω λοιπόν ότι το έγγραφο εδώ είναι τεχνικό περισσότερο. Έχουμε μιλήσει για το Frontex αλλά δεν έχουμε μιλήσει για τους ε, κώδικες που διέπουν το Schengen και την χορήγηση των θεωρήσεων. Οι συστάσεις μας είναι πιο περιορισμένες όχι μόνο γιατί διαφέρουμε επί της ουσίας αλλά κυρίως γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύντομα θα εκφραστεί για συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν το έγγραφο εργασίας και αναφέρομαι εδώ στον κώδικα της χορήγησης θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις έχει προτείνει νομοθετικές προτάσεις ιδιαίτερα στα πλαίσια της νέας πρότασης για την ακτοφυλακή και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα εκφραστεί και θα ακολουθήσουν νέες προτάσεις και για τον κώδικα λειτουργίας του Σέγγεν. Η ομάδα μου θα αξιολογήσει τις νέες αυτές προτάσεις, οι οποίες μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και στα πλαίσια λοιπόν της αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων ελπίζουμε να καταστεί ο κώδικας αυτός ένα ασφαλές μέσο για την κάλυψη των αναγκών των χωρών των πολιτών των χωρών ε, που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους και την γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την τεχνική της υποστήριξη τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ Σεσίλ. Συνάδελφοι, τελειώνει ο χρόνος, θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Um, and I'm going to add Mrs. Winberg got, um, and Juan Fernando and Mr. Coelho. I'm going to close the speakers list there, okay? Please don't ask for the floor because we have to finish it. Κλείνει ο κατάλογος, μην ζητάτε το λόγο γιατί 6.30 πρέπει να τελειώνουμε. Όσον αφορά τους κοιόδης, η κυρία Στίβενς πρώτα. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να μείνετε στα δύο λεπτά γιατί δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε πέρα από τις 6.30. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για αυτά τα οποία ήταν. αλλά βλέπω πως ε, θέλουν στήριξη για την έκθεσή τους, αλλά πρίχνοντας ε, μια ματιά βλέπω πως ε, ε, θα έπρεπε να έχουν συμπεριλάβει όλες τις ομάδες από την αρχή της ε, διαδικασίας. Και θα ήταν και το κείμενο πολύ ε, σαφέστερο. Αυτά από την ομάδα μας. Βεβαίως είχαμε κάποια αρχική επαφή αλλά μετά τίποτα και αυτό είναι κρίμα από τη δικιά μας την Σκοπιά. Λοιπόν, τώρα για το έγγραφο εργασίας της ε, ΕΑΖΟ, το οποίο το είχα εγώ ξεκινήσει και βλέπω το ξανάγραψαν τελείως οι συγγήτριες. Ε, μην με παρεξηγείτε, κάπου το βελτίωσαν κιόλας. Και όπου προσέθεσαν πληροφορίες, ε, αλλά όσον αφορά την πολιτική, πραγματικά δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο έγραψα. Προτείνονται μη ρεαλιστικές ε, λύσεις, ε, παραδείγματο χάρη την πρόταση που κάνουν για τη μεταρρυθμίση του Δουβλίνου και το μηχανισμό επανεγκατάστασης και χωρίς να υπάρχει καμία σχέση μάλιστα και να γίνεται η σύνδεση με την προστασία των εξωτερικών ε, συνόρων. Μόνο για αναδιανομή ε, μιλάνε και παρέμβαση στα ε, εσωτερικά των κρατών. Μας είπε η Θεία Μέρκελ να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες ε, και παραμένει, παραμένουν ορθάνυχτα τα εξωτερικά σύνορα και η κοινωνική πρόνοια. Είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό για τους ε, φλαμανδούς ε, ψηφοφόρους μας. Ο Τίμωθη Κέρκοπ, ο συνάδελφος στο ECR, έχει αναλάβει τον φάκελο για την επανεγκατάσταση. Ναι, επανεγκατάσταση, αλλά με αυστηρές προδιαγραφές και αφού υπάρξει περιορισμός της εισρωής. Αυτό νομίζω θα πρέπει, αυτή η κατεύθυνση ώρα θα πρέπει να κινηθεί η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, μετά τις 6.30 βεβαίως ε, σχολάνε οι Παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε το ωράριο. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Και εσύ πάντα τηρείς τα ωράρια, οπότε δεν ήταν για σένα το σχόλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τις εισηγήτριες για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει, πολύ προσεχμένη σε κάποια σημεία. Και έχω μια σειρά από ερωτήσεις ε, σημαντικές, τις οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ώστε τα έγγραφα να μην είναι απλώς μια απεικόνηση της υπάρχουσης κατάστασης με κάποιες μικρομεταρρυθμίσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα ήθελα να σταθώ σε κάποια λίγα πράγματα. Frontex ε, γίνεται οργανισμός ε, ακτοφυλακής, προστασίας των συνόρων και των ακτών. Η νέα Frontex, ο νέος Frontex που θα παρεμβαίνει χωρίς σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, πώς θα επιλύσουμε εδώ το πρόβλημα των ευθυνών ο διευθυντής του Frontex δεν είναι ερετός, ε, δεν υπάρχει λογοδοσία ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου. Πρόκειται λοιπόν για έναν οργανισμό ο οποίος θα έχει όλες τις εξουσίες, αλλά η ευθύνη θα παραμένει η ευθύνη των κρατών μελών. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά το Frontex είναι η παρεμβάση σε τρίτες χώρες χωρίς ε, επαρκή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μήπως θα έπρεπε αυτό να αναφέρεται σαφώς στην έκθεση και επίσης ε, έρευνα και διάσωση, search and rescue. Δεν ε, μου φαίνεται να είναι πλέον προτεραιότητα στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και αυτό στην έκθεση. Τελευταίο θέμα, οι τρίτες χώρες, κυρίως ε, αυτό το οποίο με ανησυχεί σήμερα είναι η Τουρκία. Μου φαίνεται σαφές ότι μία σχέση αυτής της μορφής θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι οι σχέσεις συνεργασίας μιας χώρας που ε, παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα αναστέλλονται αυτομάτως. Ε, σταματάω γιατί είμαι στα 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριες. Πιστεύω ότι έγινε εξαιρετική δουλειά. Το έγγραφο εργασίας είναι εξαιρετικό στο τμήμα που αφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Σύλλου. Για τα άλλα δύο όμως ε, έχω αμφιβολίες αντίστοιχες με αυτές που ανέφερε προηγουμένως η Μπάρμπαρα Σπινάλη ότι έχουμε έναν απολογισμό της κατάστασης, αλλά όσον αφορά τις προτάσεις ε, λείπουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν και δεν είναι σε καμία περίπτωση σαφή. Όσον αφορά τώρα το σύστημα ασύλου, σίγουρα είμαι υπέρ ε, του εγγράφου. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές ε, τη σπάση ότι το σύστημα του Δουβλίνου είναι πλέον παροχημένο και θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Με κάποιες ενοχές ε, και με μεγάλη καθυστέρηση το αντιλήφθηκαν οι περισσότεροι, επομένως πρέπει να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση από την οποία επικρεμάται η όλη έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα κεντρικό για την ε, καταγραφή και επεξεργασία των αιτήματων ασύλου. Σε αυτό συμφωνώ, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε και κάποιες ε, ε, μετακινήσεις σε δεύτερο στάδιο. Νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων είναι εδώ ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Υπάρχει πρόταση για μια θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους. Ε, νομίζω ότι και με αυτό συμφωνώ. Επειδή τελειώνει ο χρόνος και είναι πολλά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους και θα έχουμε χρόνο να τα ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον. Λυπάμαι που μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκθεση. Πρέπει να πούμε τόσα πολλά πράγματα και το χρονοδιάγραμμα δεν ε, ήταν πάρα πολύ καλό και όλα τα υπόλοιπα έχουν καθυστερήσει. Να προχωρήσουμε. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Δύο λεπτά συνάδελφοι γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κοράου για αυτό το οποίο μόλις είπε. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ακούσαμε λοιπόν τις εισηγήτριες ε, και την κυρία Κιέγγε και γίνεται εδώ πέρα αρητή αναφορά στην ε, σημασία του να ανοίξουν νόμιμες ε, δίωδοι για τους ετούντες άσυλο που προσπαθούν να χτυπήσουν την πόρτα, τις πύλες της Ευρώπης. Εγώ είμαι εξάλλου και εισηγητής του κώδικα βίζας και αυτό το οποίο προσπαθώ να πω για τις ομάδες ακόμα που ακόμα δεν το θέλουν είναι ακριβώς αυτό. Ε, να δεχτούμε ανθρωπιστικές βίζες. Όχι μόνο για να υπάρχει συνέπεια με άρθρα 19 και 25 για τον κώδικα θεωρήσεων αλλά και για να ανοίξει μία νόμιμη δίωδος για όσους θέλουν να ζητήσουν ανθρωπιστική βίζα με βάση το δεσμευτικό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κράτους μέλους. Ευχαριστώ λοιπόν την προσοχή και των εισηγητών και των πολιτικών ομάδων το στο ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτό το εξαίρετο έργο με τα όσα θα γίνουν στον κώδικα θεωρήσεων. Ευχαριστώ Κόλιο. Να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, συναδέλφους μας για τη δουλειά που έκαναν. Να αναφερθώ τώρα στη διαχείριση των συνόρων και την βίζα. Ειδικά η διαχείριση των συνόρων καθιστά σαφές πω δεν υπάρχει μια μαγική λύση για το θέμα αυτό. Ποιος ο στόχος καλύτερης διαχείρισης συνόρων εάν ε, δεν έχουμε ένα σύστημα ασύλου που λειτουργεί ή δεν υπάρχει συνεργασία με τρίτες χώρες. Πρέπει να έχουμε μια συνολική. Βλέπουμε εδώ πέρα από το έγγραφο αυτό πως η διαχείριση των συνόρων βασίζεται σε δύο αρχές που επίσης ε, είναι βάση της, ε, βάσης, ε, της περιοχής εγγενία αμοιβή εμπιστοσύνη και η κοινή ευθύνη. Βλέπουμε λοιπόν πως αφενός ο πυλώνας είναι αμοιβία εμπιστοσύνη, απ' την άλλη η Frontex είναι μέρος της κοινή ευθύνης καθώς όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά ακριβώς την ανάλυση κινδύνου και διαχείριση των συνόρων. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε το τι θέμε από την Σέγγεν και αυτό θα συζητήσουμε αύριο το πρωί, όμως δεν θα αναφερθώ τώρα. Επανέρχομαι στις ε, προηγούμενες παρατηρήσεις μου. Δεν είναι μαγική η λύση, αλλά αν είναι να παραμείνει ολόκληρη η ζώνη Σέγγεν και να καλωσορίζουμε όσους αναζητούν άσυλο στις ακτές μας, χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Όχι μόνο, αλλά και χρειαζόμαστε λοιπόν αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή ανάληψη ευθυνών. Εγώ καλωσορίζω την πρόταση για κοινή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Το Κοινοβούλιο δικαίως αναζητά μια στρατηγική που θα καλύπτει όλα τα στοιχεία. Χρειάζεται να συνεχίσουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και στα μέτρα που υπάρχουν ήδη Σε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σούνιμπερν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω ότι έχουμε κάποιες αδυναμίες στην προστασία των σύνορων και κάποιες χώρες παίζουν τον ρόλο ε, διαμετακόμισης, κέντρων διαμετακόμισης. Στην Ιταλία και στην Ελλάδα το σύστημα δεν δουλεύει όμως καλά. Τι γίνεται για την υποδοχή όλων αυτών των ανθρώπων τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε και του χρόνου να έχουμε 2-3 εκατομμύρια ανθρώπων που θα έλθουν από τα ίδια κανάλια. Γιατί έχουμε φυσικά και τους οικονομικούς μετανάστες πέρα από τους πρόσφυγες. Μέχρι τώρα μόνο 160 άνθρωποι έχουν επανεγκατασταθεί. Λοιπόν δεν είναι η κατάσταση καλή. Αυτές οι ποσοστώσεις οι οποίες έχουν αποφασιστεί, γιατί δεν έχουν προχωρήσει, τι συνέπειες θα υπάρξουν για τις χώρες που δεν υποδέχονται τους αριθμούς που έχουν αποδεχθεί. Θα υπάρξουν κυρώσεις, θα τους πούμε απλά να είναι έτοιμοι για του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στις εισηγήτριες. Σύντομες παρακαλώ. να σας ευχαριστήσω όλους για τις ε, δηλώσεις σας. Θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση σε βάθος στο μέλλον. Απαντώ μόνο στην κυρία Σπινέλη για τη νέα υπηρεσία και για τις αλλαγές στο Frontex σχετικά με την πρόταση κανονισμού. Το Search and Rescue είναι βασική προτεραιότητα για μας. Είναι σημαντικό κομμάτι του συστήματος διαχείρισης των συνόρων δεν θα μακρηγορήσω, σας ευχαριστώ πάντως όλους και εύχομαι καλές γιορτές. Ευχαριστώ Κλοντ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και την Τσετσίλια φυσικά. Ελπίζω ότι τα έγγραφα αυτά είναι καλογραμμένα και ελπίζω να μπορέσουν να εφαρμοστούν επί της ουσίας με πολυκομματική στήριξη. Ευχαριστώ τους Κιώδης επίσης για τη συνεισφορά τους να απαντήσω σε αυτά που είπε η Στίβενς. Κάποια από τα θέματα τα οποία έθεσε έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλα έγγραφα εργασίας και θα συζητηθούν εκ νέου όταν φτάσουμε στην τελική έκθεση. Βλέπω τις τροπολογίες, θα εξετάσω τις τροπολογίες και ελπίζω να υπάρξει μια απεραιτέρω επαφή και συζήτηση πριν καταλήξουμε στο έγγραφο το οποίο θα ε, φτάσει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι η δουλειά σας δεν είναι πάρα πολύ ε, εύκολη γιατί την ώρα που διαμορφώνεται το κείμενό σας έρχονται συνέχεια νέες προτάσεις, ακούγονται νέες προτάσεις, άγραφες κάποιες από αυτές ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πετύχει κανείς ε, σε μια κινούμενη κατάσταση την απαιτούμενη συνένεση. αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και ευχαριστώ τις εισηγήτριες για την καλή δουλειά και ελπίζω ότι στις 18 του μηνός θα έχουμε ένα πρώτο κείμενο και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σε αυτό με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Σας ευχαριστώ όλους. Θα τα πούμε αύριο στις 9. Όσους από σας είστε εδώ. Αλλιώς χρόνια πολλά αλλά πρέπει να είστε εδώ αύριο στις 9 γιατί αλλιώς θα νιώσω μοναξιά